Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε. συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχετε το... την πρόταση να μην ψηφίσουμε σήμερα την ε, γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή, να το αναβάλουμε για αύριο. Αν συμφωνείτε, σήμερα θα ψηφίσουμε απλά για την έκθεση για την ε, απαλλαγή δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Οπότε συμφωνούμε. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε πρώτα απ' όλα την, το ηλεκτρονικό σύστημα. Ελπίζω να έχετε τις κάρτες μαζί σας για να ξεκινήσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ωραία. Ξεκινάμε. Λοιπόν, παράγραφος 1 Τροπολογία 5, μέρος πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μέρος δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 7 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά εποχέ. να το επαληθεύσουμε τροπολογία 8 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά εποχέ. δεν είναι σαφές να το επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή καταπίπτει 13 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφεται. τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 16 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. αποχέ Απορρίπτεται. Να παλαιθεύσουμε το πρώτο μέρος τροπολογίας 16 είπε Ε, άρχιτε Πέρας. Δεκτή, μάλιστα. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή, σαφώς. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Να το επαληθεύσουμε. Την 17. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή τοπολογία 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τοπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή τοπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τοπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ. Κατά αποχές Τώρα η έκθεση στο σύνολό τη με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Σας ευχαριστώ. Συγχαίρω τον Σίγητη. Ευχαριστώ όλους όσους ε, δούλεψαν και ειδικά τη γραμματεία. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίζω τον Επίτροπο, τον κύριο Σέμετα. Καλώς ήρθατε. Συχνά έρχεστε στην Επιτροπή μας, αλλά σήμερα θα συζητήσουμε την Επιτροπή διαδικασία απαλλαγής. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη και δίνουμε τον λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. ήθελα λοιπόν να ακούσουμε την εισαγωγή για το τμήμα αυτό του προπολογισμού. Κυρία Καλιονάιτη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε Σεμέτα. Στι επαφέ που είχαμε και στι ακροάσει που γίνανε στο παρελθόν, είχαμε τη δυνατότητα να συνημερώσουμε περισσότερο για την ετήσια έκθεση του 2012 από το Ελεκτικό Συνέδριο. Θα επικεντρωθώ σήμερα στο πρώτο κεφάλαιο τη έκθεση αυτή και θα μα δοθεί έτσι η δυνατότητα να συζητήσουμε περισσότερο τι επιπτώσει όσον αφορά την κατανάλωση και τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Ποιε είναι οι αλλαγέ που έχουμε το 2011. Η γενικότερη εικόνα ομοιάζει με πέρυσι και αυτό φαίνεται στην δήλωση αξιοπιστίας του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η δήλωση αξιοπιστίας ε, παρέχει μια γνωμοδότηση όσον αφορά τους λογαριασμούς, καθώς επίσης και τρεις επιμέρους γνωμοδοτήσεις όσον αφορά την κανονικότητα των συναλλαγών και έχουμε συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις για συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς. Επίση, έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να καταλάβουμε πώ λειτουργούν οι διαφορετικές πτυχές της οικονομικής διαχείρισης Ευρωπαϊκή Ένωση. Για έκτη συνεχή φορά έχουμε από το Ελεγκτικό Συνέδριο μια έκθεση χωρί επιφυλάξει όσον αφορά τους οικονομικού λογαριασμού Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να υποβάλει ξεκάθαρες γνωμοδοτήσεις και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει και στο μέλλον ακολουθώντας τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Για άλλη μια φορά το λεκτικό συνέδριο κατέληξε ο συμπέρασμα ότι όλες οι συναλλαγές ανάληψη υποχρεώσεων δεν είχαν κανένα ουσιαστικό λάθος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασιζόμενη σε εκτιμήσει των κρατών μελών είναι σε θέση να υπολογίσει και να συλλέξει σωστά τι ενισφορέ των κρατών μελών. Η θετική αυτή γνωμοδότηση για την ανάληψη υποχρεώσεων είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ξεπεράσει τα δημοσιονομικά τη όρια κάθε φορά που υπόσχεται για τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων κοινοτικών κονδυλίων. Παρ' όλα αυτά έχουμε ουσιαστικό σφάλμα σε κάποιου τομεί. Το σφάλμα αυτό εντοπίζεται κυρίως στους λογαριασμούς του 2012 όσον αφορά τις πληρωμές που έχουν αναλυφθεί, όπου έχουμε μία αύξηση 0,9% σε σχέση με πέρυσι, 4,8% για φέτος, 3,9% για το παρελθόν έτος. Το 1 τρίτο της αύξησης αυτής έχει να κάνει με την προσέγγιση δειγματοληψίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2012 το Ελεκτικό Συνέδριο βελτίωσε το δειγματοληπτικό του μοντέλο και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε συγκεκριμένες αιτήσει κάλυψης δαπανών από τα κράτη-μέλη που εξετάζονται και καλύπτονται στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έναν ομοιόμορφο τρόπο. Κατά αυτόν τον τρόπο ακολουθούμε την λογιστική σε δουλευμένη βάση, τη μέθοδο δηλαδή αυτή, και κατά αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση όσον αφορά την κτηματολοψία. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε και πιο συγκρίσιμα δεδομένα για όλο τον κοινοτικό προπολογισμό. Το 2012 το εκτιμόμενο σφάλμα για την κοινή χρήση ήταν 5,3% σε σχέση με το 4,3% για όλους τους άλλους τρόπους ε, ε, δαπανών. Τα οικονομικά αποτελέσματα, τα αποτελέσματα ελέγχου του 2012 καταδεικνύουν ότι ε, το σφάλμα δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα μόνο τμήματα του προπολογισμού, αλλά καλύπτει πάρα πολλούς τομείς του προπολογισμού. Οι βασικοί λόγοι για το σφάλμα αυτό παραμένουν οι ίδιοι. Δεν καταφέρνουμε να τηρήσουμε όπως θα έπρεπε όλους τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων και επίσης υπάρχουν διάφορα σφάλματα που σχετίζονται με μη επιλέξιμα προγράμματα, μη επιλέξιμες δαπάνες, καθώς επίσης και σφαλμένη δήλωση δαπανών για τον αγροτικό τομέα. Έχουμε εντοπίσει τα σφάλματα αυτά πολλές φορές και στο παρελθόν και βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν στο μέγιστό του το εφιστάμενο σύστημα ελέγχων θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να συνέβαινε κάτι τέτοιο, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρναμε να, να περιορίζαμε πολύ περισσότερο τα σφάλματα τα οποία έχουμε εντοπίσει. Τώρα, όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, έχουμε τη δυνατότητα να καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε αυτοματοποιημένες οικονομικές διορθώσεις. Και αυτό θα πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον. Χάρη στη δική σας την Επιτροπή έχουμε πραγματικά πάρα πολύ καλές και συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με ένα αυτόματο σύστημα καθαρών οικονομικών διορθώσεων. Πιστεύουμε ότι αν ακολουθήσουμε το σύστημα αυτό των καθαρών οικονομικών διορθώσεων θα έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε ακόμα και τη συμπεριφορά των αρχών των κρατών μελών. Τώρα, το αν οι διατάξει αυτέ θα οδηγήσουν σε περισσότερε καθαρέ διορθώσει και πραγματικά θα διηγηθούμε σε χαμηλότερο επίπεδο σφάλματο, αυτό εξαρτάται από πάρα πολλού παράγοντε. Επί του παρόντο δεν είναι δυνατόν να υπολογίσουμε τι επιπτώσει που θα έχουμε, αν δεν γνωρίζουμε πώ το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη. Ωστόσο, ένα σημαντικό παράγοντα θα είναι η δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλων θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εντοπίσουν σημαντικέ αδυναμίε και προβλήματα που θα οδηγήσουν προφανώ σε καθαρέ ή συνέχεια οικονομικέ διορθώσει. Ας επικεντρωθώ τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλές φορές και στο παρελθόν. Τη σύνδεση, τη διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο επίπεδο σφάλματος που εκτιμά το ελεγκτικό συνέδριο και το πραγματικό ποσό οικονομικών διορθώσεων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πρόσφατη γραπτή και προφορική ανακοίνωσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν λαμβάνει υπόψη του στις οικονομικές του διορθώσεις το εκτιμόμενο ποσοστό σφάλματος και κατά αυτόν τον τρόπο δεν έχουν συμπεριληφθεί τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ε, οικονομικές διορθώσεις όπως θα έπρεπε το 2012 και δεν έχει διορθωθεί το, ποσοστό αυτό, το ποσό με συγχωρείτε αυτό, με το ποσοστό του 4,8% όσον αφορά το εκτιμόμενο σφάλμα. Οι διορθώσεις που έχουν γίνει δύο στον τομέα της συνοχής έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα 2000-2006, όπου το Ελεκτικό Συνέδριο εντόπισε υψηλότερο επίπεδο σφάλματος. Τα επίπεδα διόρθωσης σχετίζονται με την περίοδο 2000-2006 και πολλές φορές το επίπεδο σφάλματος θεωρείται ότι είναι υψηλότερο. Πολλές φορές βέβαια το επίπεδο αυτό σφάλματος θεωρείται ότι δεν έχει καμία διασύνδεση με το επίπεδο σφάλματος του 2012. Κάποιες από τις οικονομικές διορθώσεις που γίνονται για άλλους τομείς δεν σχετίζονται με σφάλματα που έχει εντοπίσει, με διορθώσει που έχει κάνει το λεκτικό συνέδριο για άλλου τομεί. Το λεκτικό συνέδριο λαμβάνει υπόψη του τι οικονομικέ διορθώσει τι οποίε εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο όμω αυτέ που έχουν οδηγήσει σε λεπτομερή διόρθωση των δαπανών ή τη αποπληρωμή κάποιων ποσών κατά τη διάρκεια του τρέχοντο έτου. Οι διορθώσει αυτέ ουσιαστικά έχουν οδηγήσει σε μείωση του εκτιμόμενου σφάλματο για το έτο 2012. Τώρα, το αν η διόρθωση έχει επίπτωση σε επίπεδο προγράμματο ή όχι, αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τη δράση που τελικά αναλαμβάνουν οι κρατικέ αρχέ, οι αρχέ των κρατών μελών. Με το εφιστάμενο σύστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τα απαραίτητα μέσα για να καταφέρει να πετύχει τι απαραίτητε αυτέ διορθώσει σε επίπεδο προγράμματο. Από την άλλη, όμω, φαίνεται το λεκτικό συνέδριο μπορεί με τη δικιά του τη στάση να επηρεάσει τη συμπεριφορά του κράτου μέλου βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή όπου έχουμε αρνηθεί να προχωρήσουμε σε μια καταποκοπήν διόρθωση οικονομική είχαμε και θετικές επιπτώσεις όσον αφορά το έτος 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θεωρεί ότι το ποσό της οικονομικής διόρθωσης κράτος μέλος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα αξιόπιστος δείκτης για το επίπεδο σφάλματος κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφό της με τίτλο «Προστασία του κοινοτικού προπολογισμού» και σύμφωνα με το σημείο παριθμών 6 που παρουσίασε στο λεκτικό συνέδριο έχει εντοπίσει συγκεκριμένα τρία κράτη-μέλη τα οποία συμβάλλουν κατά ένα ποσοστό 80% στο συνολικό επίπεδο σφάλματο. Από ό,τι φαίνεται όμως το σφάλμα έχει υψηλότερο ποσοστό από αυτό το οποίο έχει εκτιμήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε ποιες διορθώσεις έχουν γίνει σε προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού, αλλά ακόμα και αν ληφθεί αυτό υπόψη, δεν θα έχουμε την πλήρη σφαιρική εικόνα όσον αφορά το επίπεδο σφάλματο. Τέλος, το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις αιτήσει πληρωμών. Ξέρετε ότι το ίδιο είχαμε δει και το 2013. Η γενικότερη πίεση στον κοινοτικό προπολογισμό αντικατοπτρίζεται από τα αυξανόμενα ποσά τα οποία κρεμούν όσον αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίση να καταφέρει να αντιμετωπίσει όλε αυτέ τι αναλήψει υποχρεώσεων για συγκεκριμένε πληρωμέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα κρεμή ζητήματα πληρωμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει ε, σε ένα ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να βρεθεί ένα νέο τρόπο για να εξασφαλιστεί η ταμιακή ροή όσον αφορά τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσά και την Επιτροπή σα για τον επικοδομητικό διάλογο και συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια τη διαδικασία απαλλαγή του 2012. Να ευχαριστήσω επίση και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και την συμβολή τη της δικής της Επιτροπής, προκειμένου να καταφέρουμε να βελτιώσουμε το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλιουλάιτ, εξ ονόματος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Τώρα το λόγο έχει ο Πίτροπος Σεμέτα. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ισηγητά, ισότιμοι βουλευτές και μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Αυτή η ακρόαση σήμερα γίνεται μετά από μια σειρά επαφών που είχατε με τους συναδέλφους επιτρόπους που έχουν αναλάβει σημαντικές πολιτικές και σε σχέση με τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις τις τόσο σημαντικές από τότε που είχαμε ε, την ετήσια έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου τον Νοέμβριο. Εγώ και οι υπηρεσίε μα έχουμε στενή επαφή με την Επιτροπή σα και πιστεύω ότι τώρα θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα τα οποία διακυβεύονται και αυτή η διαδικασία τη ε, απαλλαγή μπορεί να βοηθήσει όλου του εμπλεκομένου και τα κρατημέλη, ούτω ώστε να βρεθεί ο καλύτερο τρόπο για μια χρηστή και υγιή ε, δημοσιονομική διαχείριση του προπολογισμού. Μια νέα περίοδο προγραμματισμού σημαίνει νέου κανόνε, νέα εργαλεία, νέε διαδικασίε που αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να μειώσουμε περαιτέρω ε, τον ε, κίνδυνο ασφάλματο και να μπορέσουμε να έχουμε την προσθέμενη αξία που προσδοκούμε με τρόπο που διακρίνεται από διαφάνεια και καλή σχέση κόστο αποτελέσματο. Για να δούμε τώρα την ετήσια έκθεση. Με μεγάλη μου ικανοποίηση διαπιστώνω ότι το ενεργό Συνέδριο ενέκρινε του λογαριασμού, τον ισολογισμό ούτω πίνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για έκτη φορά ε, στη σειρά, έκτη χρονιά στη σειρά και με αυτόν τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι οι υποχρεώσει, ε, έσοδα και δαπάνε δεν έχουν ουσιαστικά λάθη και επομένω ε, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα για αυτέ τι συστάσει και να δεσμευτούμε να κάνουμε την υλοποίηση, να προσθέτουμε την υλοποίηση όσο γίνεται για να μην έχουμε πλέον τέτοια λάθη για αυτά που έχουν επισημανθεί. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε τώρα κάποιες επιμέρους εκθέσεις για, σε σχέση με τις συστάσεις που έχουν διατυπωθεί και με την Επιτροπή τη πρόοδου του οικονομικού ελέγχου. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Ότμπο, εδώ που βρίσκεται δίπλα μου, να βελτιώσουμε περαιτέρω την εποπτεία που αναλαμβάνουν οι υπηρεσίε μα και να μπορέσουμε να διευκολύνουμε το συνέδριο σε σχέση με τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν και τις ε, ε, επιπτώσει του Κάθε τον τρόπο θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποια προγραμματά δράσης τα οποία πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα, να είναι προσβάσιμα στο ελληνικό συνέδριο, να μπορέσουμε έτσι να, σχολιάσουμε ή να έχουμε μια κοινή γλώσσα και επίσης να μπορέσουμε να ιεραρχήσουμε τις σχετικές ε, συστάσεις. Οπότε παρά την ε, αποτελεσματική υλοποίηση των συστάσεων του συνεδρίου θα πρέπει να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας, διότι έχουμε τον ε, βαθμό σφάλματος από το 3,9 το 2011, το 2012 4,8 και όπως ξέρετε το έντριτο αυτής της αύξησης ε, οφείλεται στην καινούρια δημοτελεπτική μέθοδο του συνεδρίου. Όσον αφορά τις άμεσες δαπάνες, πέραν αυτού έχουμε αυτές τις ε, φάπεξ κατά διορθώσεις, οι οποίες έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν η οι αξιώσεις πληρωμών έχουν ληφθεί υπόψη από το συνέδριο, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι και του 2012 το σφάλμα ευθυγραμμίζεται με τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την κοινή διαχείριση, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δυναμικό τρόπο προσπαθεί να διερευνήσει τις πηγές αιτίες των σφαλμάτων ε, σε συνεργασία με τα κρατή-μέλη και εστιάζει τις προσπάθειες στα πιο ρυψογίνδυνα ε, προγράμματα σε σχέση με τα κράτη-μέλη που δεν έχουν τόσο καλές επιδόσεις για να μπορέσουμε να έχουμε επομένω μια τέτοια αποτελεσματική διαχείριση, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις δομές, όσον αφορά τις κατευθυντήριες προς τους δικαιούχους της πολιτικής ε, συνοχής και γι' αυτό ε, εμπορσταθούμε να έχουμε κάποιες δράσεις εκπαίδευσης προς τους εθνικούς ελεγκτές αλλά και προς τους δικαιούχους. Επίσης, έχουμε ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να απλουστεύσουν τις ε, επιλογές κόστος, όπως γνωρίζετε. Δεν διαπιστώσαμε σφάλματα στο 26% ε, του ESF σε σχέση με αυτές τις απλουστεύσεις, τη δε περιφερειακή πολιτική, εστιάσαμε την προσοχή μας στην αξιοπιστία των ε, ε, ελέγχων από τις ε, αρμόδιες αρχές τέλος του 2013 η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής είχε καλύψει 47 περιφερειακά ταμεία και ταμεία συνοχής σε σχέση με τις ελληνικές αρχές και είχαμε καταλήξει το 96% του προπολογισμού για τα δύο αυτά ταμεία και τα αποτελέσματα ήταν θετικά κατά τα άλλα. Τα προγράμματα δράση είχαν συγκροτηθεί και είχαμε διακόψει πληρωμές εκεί που χρειαζόταν, είχαμε βρει τι αδυναμίε και είχαμε τονίσει το, τα δύο τρίτα των, των διαδικασιών διακοπής του 2013 είχαν βασιστεί σε εθνικού ελέγχου για την γεωργία είχαμε πει ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα με τους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων, είχαμε αναλάβει συγκεκριμένη δράση σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, είχαμε πει ότι υποχρεούνται να μας κοινοποιήσουν τις ενέργειες που αναλαμβάνουν, οπότε και με αυτή τη μέθοδο είχαμε συγκεκριμένες μεταβολές, είχαμε επίσης ε, την ακύρωση ε, κάποιων προγραμμάτων υποστήριξης, αλλαγές στη διαδικασία ελέγχου και συνεργαζόμαστε και βοηθούμε τα κράτη-μέλη, αλλά ε, δεν θα ε, εμπιστευόμαστε τυφλά ε, χάρη στις αυξημένους οικονομικούς ελέγχους του Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλο ένα και περισσότερο μπορούμε να επισημάνουμε τις αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματα των εθνικών ελέγχων. Επ' αυτές τις βάσεις έχουμε κάποιο είδους πίνακες κινδύνου για κάθε πρόγραμμα το οποίο το ενημερώνουμε επί τη βάση των ε, οικονομικών ελέγχων, των ε, γενικών διευθύνσεων, των εξωτερικών ελεγκτών και ε, έτσι έχουμε την γενική έκθεση ετησίου ελέγχου. Και επομένως όταν καταρτίζουμε τα, τα μνημόνια προγραμματισμού έχουμε και προγράμματα οικονομικού ελέγχου Οπότε μπορούμε να επισημαίνουμε ε, πού υπάρχουν τα δυνατά σημεία στα ε, προγράμματα τα οποία εφίστανται περισσότερου κινδύνου με αυτή τη μεθοδολογία. Επίση, μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματική κατανομή ε, των ελεγκτών μα και έτσι μπορούμε να βλέπουμε σε σχέση με την επίδοση κάθε κράτου μέλου που υπάρχουν μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Ο, όποτε έχουμε καλέ επιδόσει από τα κράτη-μέλη, αυτά τα κράτη-μέλη και περιφέρειε ε, υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς ελέγχους ε, και το αντίθετο. Άπαξ και επισημάνουμε σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση και στους ελέγχους κάποιου κράτους μέλους. Σταματούμε τις πληρωμές προς το συγκεκριμένο κράτος μέλος το 2012 δε διακοπές ε, όσον αφορά κάποια ταμεία για αληθική πολιτική, κοινωνική, συνοχής, περιφερειακή έφτασαν αυτές τις διακοπές τα 5 δις ευρώ και ενώ το 2011 ήταν το αντίστοιχο πόσο 2,6 δις ευρώ. Ε, οπότε, όποτε είχαμε κάποια λάθη, δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να έχουμε αυτά τα διαφορετικά μέτρα και όπως εξήγησα σε μια πρόσφατη ανακοίνωση για τον προϋπολογισμό, οι διορθώσεις και οι ανακτήσεις έχουν σημαντικά αυξηθεί. Φτάσαν τα 4,4 δις ευρώ το 2012 σε σχέση με το 1,8 δις το 2011 για την περίοδο 2009-2012 αυτά τα διορθωτικά μέτρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 2% του συνόλου των πληρωμών. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον ρυθμό σφάλματος των ετήσιων με τον πολιετή διορθωτικό μηχανισμό θεωρούμε ότι ε, ο ρυθμός, ε, το ποσό των σφαλμάτων αυτά τελικού τελικούς δικαιούχους και αυτό όμως δεν μπορεί να είναι η μόνη ένδειξη για να μπορέσουμε να κρίνουμε τι γίνεται τις περιπτώσεις της συνδιαχείρισης όσον αφορά τις επιδόσεις του κάθε κράτους μέλους. Όλα αυτά πρέπει να τονίσουμε ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, η προστασία των ε, φορολογουμένων των συμφερόντων του σε εθνικό επίπεδο πρώτα-πρώτα ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτοί κύριοι βουλευτέ, εμεί συμφωνούμε με την άποψη του Συμβουλίου ότι η έναρξη τη καινούργια δημοσιονομική περίοδου θα πρέπει να είναι αφορμή, ούτω ώστε να αναβαθμιστεί ο υποπτικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να έχουμε τον ε, καλύτερο δυνατό τρόπο χρήση του προστασίου μας για να μπορέσουμε να διορθώσουμε, να μπορέσουμε να προλάβουμε σαν ε, συνομοθέτε. Ε, άμεσα αντιδράσαμε στην επιστολή σας προς τον πρόεδρο Μπαρόσο και 13 2013 είχαμε αυτή την ανακοίνωση για τις καθαρές δημιουργικές διορθώσεις και όπως έγινε και στη Γεωργία τα κράτη-μέλη οπωσδήποτε πρόκειται να απολέσουν ε, πόρους στην πολιτική συνοχή εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ελεκτροσυνέδριο Συνέδριο επισημάνει σημαντικές αδυναμίες που θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί από τις εθνικές αρχές. Η ιδέα διαδικασία η οποία ενεργοποιεί αυτές τις ε, καθαρέ διορθώσεις είναι συστηματική. Και αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζεται χωρίς ε, κάποιου είδους ε, ε, διακριτική επιλογή και βασίζεται σε αντικειμενικά και διάφορα κριτήρια. Στη Φιλανδία το Μάιο του 2011 με ελέγχους διαπιστώσαμε ότι το συνολικό σύστημα ελέγχου ήταν αποτελεσματικό εκτός σε σχέση με κάποιες διατάξεις, κάποιες προϋποθέσεις ε, αγοράς ε, εξοπλισμού που δεν διαπόντουσαν από πάρα πολύ σωστούς ελέγχους ε, και δεν είχαν οριστεί σωστά. Επίσης βρήκαμε κάποια λάθη που αντιστοιχούν στο 2,7 των πληρωμών που σημαίνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε πρόκειται η Φινλανδία να πληρώσει και πάλι πίσω στον προϋπολογισμό του 2014 κάτι το οποίο θα θεωρηθεί έσοδο. Αυτό σημαίνει ότι ε, αυτή είναι μία από τις 147 ε, διορθώσεις της αγροτικής ε, πολιτικής του 2013 που αντιστοιχούν σε 1,1 ε, δις ευρώ. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι οι καθαρές διορθώσεις αποτελούν ένα τρόπο που είναι σαν τελευταία λύση και οπότε θα πρέπει να δούμε ότι αυτό βοηθά να επηρεάσουμε την συμπεριφορά των κρατομελών που δεν έχουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να καταστήσουμε υπεύθυνα τα κράτη-μέλη. Να έχουμε δηλώσεις διαχείρισης από τις εθνικές αρχές, κάτι το οποίο υπόσχεται πολλά. Επίσης, ε, αυτές τις δηλώσεις θα πρέπει να τις ε, ε, συνοδεύουν κάποιες πληροφορίες που θα πρέπει να είναι πλήρες, να είναι αξιόπιστες και κατά αυτόν τον τρόπο θα ε, έχουμε ε, μία ανεξάρτητη γνώμη ελεγκτού για το τι κάνουν τα μελη Παρ' όλα αυτά, συμφωνούμε με το Κοινοβουλίο Συναφορά, αφορά την προσθέμενη αξία των ε, εκουσίων εθελοντικών, εθελουσίων, εθνικών δηλώσεων σε πολιτικό επίπεδο, οπότε έτσι πρόκειται να αναβαθμίσουμε την υπευθυνότητα και και την λογοδοσία των μελών που διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά χρήματα. Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διοργανική και έδωσε την έμεινευση ο Γιάν Μίλτερ έχει αναλάβει τα καθηκοντά της και θα πρόκειται πάρα πολύ σύντομα να έχουμε ε, κάποια δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δύο πρώτων συναντήσεων. Επίσης έχουμε ένα καινούριο πλαίσιο, αυτό δείχνει τι πρόκειται να γίνει με την προσθέμενη αξία ε, που αφορά τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιχειρήσεις και τους Ευρωπαίους. Και επίσης θα έχουμε συγκεκριμένους στόχους, θα έχουμε επίσης δείκτες ε, για πάρα πολύ σημαντικά σημεία όσον αφορά τις επιδόσεις και οπότε ε, έτσι θα έχουμε εκθέσεις για την πρόοδο και θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα σημαντικά ορόσημα, κάποιες διάμεσες ε, αναθεωρήσεις και όπου χρειάζεται πρόκειται να προσαρμόσουμε τα προγράμματα. Οπότε, φυσικά και οι ειδικέ εκθέσεις ε, των, του, του, του, του Ελληνικού Συνεδρίου είναι πάρα πολύ πολύτιμες και θα πρέπει επομένως να τις λάβουμε υπόψη για τις προτεραιότητές μας. Εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι συμφέρον μας να εξασφαλίσουμε ότι εκτελείται ο ευρωπαϊκός μενουσιακός τέλο πάντων προπολογισμό σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η απαλλαγή για τη χρήση του 2012 επομένω είναι η καλύτερη ευκαιρία που υπάρχει ούτω ώστε να προωθήσουμε την καλύτερη υλοποίηση του νέου ε, πλαισίου. Θα συνεχίσουμε το έργο μας σε στενή συνεργασία με τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, ώστε να έχουμε μια σωστή προσέγγιση για την νέα προγραμματική περίοδο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Σαμέτα, κύριε πίτρο, κύριε Πρόεδρος. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή των απαλλαγών φέτος. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ κύριε Καλιουλάιντ για αυτά τα οποία μας είπατε. Έχουμε Λοιπόν, μια σειρά εδώ πέρα πραγμάτων που είναι αποφασιστική σημασίας για την αξιολόγησή μας, βεβαίως η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά και αυτά τα οποία μας είχε πει ο Γκάιερ, ο κύριος Γκάιερ στην τελευταία του έκθεση για τον κοινοτικό προπολογισμό, αποτελούν σημαντική βάση και τώρα έχουμε άλλη μια βάση την ανακοίνωση της Κομισιόν για τις ε, δημοσιονομικές διορθώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για το ότι ανταποκριθήκατε στην πρωτοβουλία που είχαμε και μας δώσετε μια καλή βάση εργασίας. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ σε κάποια πράγματα για να αξιολογήσουμε συνολικά τα τρία έγγραφα. Το ένα είναι η συζήτηση για το ποσοστό σφάλματος που επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Ως προς αυτό μια παρατήρηση μόνο για αυτά τα οποία είπε σήμερα ο κ. Πετροπός πως έπρεπε να μειωθεί ξανά στο 3,2%. Βεβαίω τα περισσότερα από αυτά τα ποσά δεν πάνε πίσω στο κοινοτικό προπολογισμό, αλλά ξαναχρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Και το δεύτερο επιχείρημα είναι πως μόνο 1% των διορθώσεων είναι καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις. Οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και υπάρχει και ένα τρίτο σκέλος ότι δηλαδή αυτά δεν εγγράφονται στο οικονομικό έτος ε, της διαδικασίας απαλλαγής. Γιατί άμα θέλει κανείς να είναι κακός, εάν πάρουμε το έτος 2012 και έχουμε διορθώσεις από το 2002 έως το 2006, με τις οποίες, ε, τις οποίες συνυπολογίζουμε, θα έχουμε και θετικό ε, ποσοστό διορθώσεων. Οπότε δεν στέκει αυτό, καταλαβαίνετε. Το γεγονός είναι πως για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχουμε λοιπόν μια αύξηση, οπότε είναι αρνητική αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα επίση να αναφερθώ συγκεκριμένα και στις καθαρέ δημοσιονομικές διορθώσεις ε, που έχουμε τώρα μπροστά μας. Και πρέπει να πω πως πραγματικά έχουμε κάποιους νομίζω που είχαμε κάποια καινοτομία θα έλεγα, κάτι το οποίο απαιτείται γιατί η Κομισιόν γνωρίζει πως ε, η Προεδρία έχει δεσμευτεί, ο κύριος Μπαρόζο έχει δεσμευτεί προσωπικά να έχουμε κάποια μια θετική αξιολόγηση. Κάτι το οποίο δεν βλέπω να συμβαίνει. Αυτό το οποίο είναι θετικό είναι πως ε, το μέσο αυτό των καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων έχει παφείς κανόνες ε, οι οποίοι ακολουθούνται αλλά οι σαφείς αυτοί κανόνες δεν είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε αυτοματισμό και αυτό το οποίο ζητήσαμε δηλαδή. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία ζητήσαμε και δεν έχουμε. Στην δε γεωργική πολιτική τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου όσον αφορά τις καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις και για το πολύ απαιτητικό δε χρονοδιάγραμμα που θέλετε να μειώσετε στα δύο χρόνια νομίζω πως αντιβαίνει με τους εσωτερικούς στόχους που έχει θέσει η Κομισιόν ότι θέλετε εσωτερικά ε, να ε, υπάρχει μια διαδικασία 645 ημερών για την επίλυση των διαφορών. Ε, άμα εσωτερικά ο στόχος της Κομισιόν είναι ήδη τόσο γενναιόδωρος, τι να περιμένουμε τότε. Δεν βλέπω κάποια εντατικοποίηση της διαδικασίας, φοβάμαι πως θα μείνουμε στα ίδια και στα ίδια. Θα ήθελα τώρα για το θέμα της συνοχής να πω κάποια πράγματα. Εκεί όντως έχουμε τις ε, μεγαλύτερες αλλαγές. Και αυτό το οποίο πραγματικά δεν μας ευχαριστεί είναι το γεγονός πως όταν τα κράτη-μέλη ε, μέχρι τις 15 Δευτέρου που πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφα να καλύψουν κάποια λάθη μπορούν να αντικαταστήσουν χωρίς κανένα όριο τα έργα τα οποία από μόνα τους ανακάλυψαν ότι έχουν σφάλματα. Οπότε μπορούν να έχουν κάποια άλλα έργα και, και εδώ πέρα πάλι δεν υπάρχει όριο. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο οδηγεί σε μπλοκάρισμα και σπατάλει τελικά των κονδυλίων του προπολογισμού. Εμεί θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στη διαδικασία αυτή. Και αυτό επίσης το οποίο δεν ε, αντιλαμβάνομαι είναι η άμεση αυτή ε, εξέταση. Τι κάνει δηλαδή η Κομισιόν πριν από τις 15 Δευτέρου όσον αφορά τον άμεσο έλεγχο των κρατών μελών. Αυτό δεν ε, είναι αντιληπτό ούτε από τους αριθμούς ούτε από την ένταση των ελέγχων. Αυτό που είναι αντιληπτό είναι το τι κάνετε μετά τις 15 Δευτέρου όταν λαμβάνετε τα έγγραφα και η προσέγγιση ε, με βάση τον κίνδυνο που ακολουθούνται είναι πραγματικά εξαιρετική. Αυτό θέλουμε. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Η βασική διαπίστωση, αν θέλετε. Έχουμε 50 έως 60% τα κράτη-μέλη που θα έπρεπε να έχουν ανακαλύψει τα σφάλματα. Αλλά η Κομισιόν κατά βάση βασίζεται 100% στα κράτη-μέλη για την εξέταση των εγγράφων και μετά ακολουθεί των δικαιολογητικών και μετά ακολουθεί η διαδικασία που καταλήγει στη δημοσιονομική διόρθωση. Το βασικό λοιπόν για μένα είναι γιατί δεν υπάρχει άμεσος πρωτογενής στατιστικός έλεγχος, πρωτοβάθμιος στατιστικός έλεγχος των κρατών μελών χωρίς να εμπλακούν οι εθνικές ε, ελεγκτικές αρχές. Άμεσα να μπείτε στους δικαιούχους ή κομισιόν και μάλιστα να ψάξετε ειδικά τα μαύρα πρόβατα της διαρθρωτικής και της γεωργικής πολιτικής. Έτσι. Και με κάποιο αυτοματισμό. Όσο χειρότερα τα πάει μια χώρα, τόσο πιο πολύ να μπαίνει άμεσα η Κομισιόν χωρίς να εμπλέκει τις εθνικές ελεκτικές αρχές. Αυτό θα περιμέναμε εμείς και θεωρώ πως εντάξει, έχετε κάνει κάποιες καλές προτάσεις τώρα για τις ε, καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις αλλά εξακολουθεί ε, λίγο πολύ να μην χρησιμοποιεί η Κομισιόν αυτό το μέσο. Θα ήθελα να πω κάτι τώρα για το τι γίνεται όταν ανακαλύψετε κάτι μετά τις 15 Δευτέρου. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια διαδικασία έχετε. Βλέπω τυχαία πράγματα. Ε, θα θέλαμε κάποια διαφάνεια. Αλλά το ότι όταν μιλάτε για σοβαρές ελλείψεις και εδώ πέρα η έμφαση είναι στη λέξη σοβαρές και μόνο τότε προχωράτε σε διορθώσεις. Δεν το ορίζετε αυτό. Τι είναι η σοβαρή ε, έλλειψη. Υπάρχει κάποιο ε, χρηματικό όριο, ένα κατόφλι και μετά υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι και άλλο ένα παραθυράκι για τα κράτη-μέλη. Μπορούν δηλαδή να δηλώσουν και μετά τις 15 Δευτέρου. Μέχρι δηλαδή να ξεκινήσει την έρευνα το, η, η Κομισιόν μπορεί να δίνει στοιχεία το κράτος μέλος για να καταστεί δυνατή η αντικατάσταση των έργων. Και αυτό παραθυράκι. Δηλαδή, εάν ακολουθούσαμε καθαρά την διαδικασία την οποία περιγράψετε πάρα πολύ καλά, όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να ελέγχουν άμεσα τα κράτη-μέλη ε, έχουν τόσα πολλά παραθυράκια ώστε φοβάμαι πως το μέσο αυτό των δημοσιονομικών διορθώσεων δεν μπορεί να να χρησιμοποιηθεί. Και δεν τηρείται αυτά τα οποία έχετε ορίσει δηλαδή. Να τα ξαναπώ λοιπόν. Η διαδικασία που βασίζεται στις εθνικές εκθέσεις και σε αυτά τα οποία βρίσκουν τα κράτη-μέλη είναι καλή, αλλά εμείς θα θέλαμε άμεσο έλεγχο στα κράτη-μέλη που ε, είναι ας πω υπότροπα και ε, χωρίς την εμπλοκή των εθνικών ε, ελεγκτικών ε, αρχών. Είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα και ο συνάδελφος ο κ. Ντόιτς ήδη Βλέπω πως έχει αρχίσει να βαριέται τόση ώρα που μιλάω, αλλά τέλος πάντων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία και βεβαίω αναμένουμε και την πράξη κατεξιοδότηση που θα υποβάλλεται και εκεί πέρα αναμένουμε κάποια βελτίωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω. Και ευχαριστώ και τον κύριο Πίπερ Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τους υπόλοιπους συναδέλφους. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να απαντήσει κατευθείαν ο κύριος Επίτροπος στον κύριο Πίπερ. Αλλά μπορούμε βέβαια και να μαζέψουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα κομμάτι των αρμοδιοτήτων, των αρμοδιοτήτων σας που αφορά λιγότερο την απαλλαγή και περισσότερο τον Όλαφα. Εγώ έπαθα πολλά πράγματα το 2012. Έμαθα πως ε, υπάρχουν κάποιες παραβιάσεις ε, του δικαίου και η Κομισιόν είναι αδιάφορη. Αξιοσημείωτο αυτό. Οπότε το ερώτημά μου είναι τι θα γίνει με την νομική ανάλυση των υποκλοπών ε, των τηλεφωνημάτων σας ε, το ρωτήσαμε αυτό, αλλά δεν θέλω τώρα να θεωρήσω απάντηση αυτό το οποίο μας δώσατε. Μετά, νομιμότητα δραστηριοτήτων κατά πολιτών της Ένωσης. Αν δούμε την απόφαση του Μαλτέζικου Δικαστηρίου για τον ε, πρόεδρο της Όλαφ. Επίσης υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις κακοδιοίκησης στον ε, Μεσολαβητή. Ξέρετε, αν δεν κάνουμε κάτι μόνοι μας, πρέπει τουλάχιστον να επιτρέψουμε να κάνει κάποιος άλλος κάτι. Αλλά αν δω πώς διαρκεί μέχρι οι εθνικοί Βέλγοι δικαστές να λάβουν απάντηση στο ερώτημά τους για τους τρεις ε, υπαλλήλους ε, του Όλαφ, πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει θέληση για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πόσο καιρό χρειάστηκε για να απαντήσετε στο ερώτημα των Βέλγων δικαστών. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι σε θέση να κάνει μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκεί πέρα θα λάμψει η αλήθεια. Είμαι σίγουρη και είμαι σίγουρη πως και τα δικαστήρια παρά τα προσκόμματα ε, θα καταφέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά ε, εσείς γιατί κλείνετε τόσο πολύ τα μάτια για τα ιστορικά προβλήματα του Όλαφ. Ε, έχουμε και σημαντική εξέταση του προσωπικού. Αν δούμε πως ένα 28% ε, του προσωπικού θέλει να φύγει από τον Όλαφ, είναι δραματικό. Και βλέπω πως είχαν νέες δραστηριότητες στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και 57% των διευθυντών δηλώνουν πως το προσωπικό τους δεν είναι ικανό για την ε, δουλειά, πρέπει να αρχίσουν να χτυπάνε καμπανάκια και συναγερμοί για την αποτελεσματικότητα. Νομίζω πως το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να κάνει μια ειδική έκθεση, μια ενημέρωση της παλαιάς ειδική του έκθεσης. Αλλά αυτό το οποίο με ανισχύει είναι η εκοφαντική σιωπή της Κομισιόν για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Μετά. Υπάρχει ένα σημείωμα που δίνει οδηγίες για την μεταχείριση απορριφθησών ε, υποθέσεων και εδώ πέρα πάλι εκοφαντική σιωπή ε, σε όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι λίγο περίεργη η σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Γιένς Γκάια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ Ήθελα, θα ήθελα να συμφωνήσω με τα περισσότερα από αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής μας πλην ενός και γι' αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πίπερ για την ε, διαφάνεια και για τις αιτίες ε, των ε, σφαλμάτων. αλλά κάπου διαφωνώ και διαφωνώ στο ζήτημα των καθαρών διορθώσεων. Όλοι έχουμε το πρόβλημα πως η πρώτη γραμμή υπεράσπισης της νομιμότητας των δαπανών είναι τα κράτη-μέλη. Και το κάνουν και εσείς είπατε κύριε Επίτροπε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πως ε, χωρίς συνεργασία των κρατών μελών δεν μπορεί να πέσει το ποσοστό του σφάλματος και θεωρώ πως οι μειώσεις αυτές να μπορούσαν ίσως να έχουν άλλο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε τα κράτη-μέλη και να υπάρχει, αν θέλετε, μια στρατηγική μαστιγίου και καρότου. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε το εξής θα μπορείτε να λάβετε τα λεφτά αν βρείτε μόνοι σας το λάθος και ναι βεβαίως πρέπει να υπάρχουν τα έργα αλλά θέλουμε να ρέει το χρήμα για να επιτύχουμε τους πολιτικούς μας στόχους. Και καλό θα ήταν νομίζω και τα κράτη-μέλη να έχουν ε, περισσότερα έργα τα οποία βεβαίως είναι άξια χρηματοδότησης. Αλλά εάν βρίσκει το σφάλμα το ελεγκτικό συνέδριο ή οι ελεγκτές της Κομισιόν, εκεί πέρα νομίζω πως ε, είναι η σειρά του μαστιγίου και πρέπει να πούμε, εντάξει, αν δεν είστε σε θέση να βρείτε τα λάθη, ε, δεν θα λάβετε τα χρήματα και βεβαίως να δούμε μετά. Αν ε, τα χρήματα αυτά δεν πάνε στο κράτος μέλος αλλά στον προπολογισμό της Ένωσης πρέπει να ξέρουμε και τι θα τα κάνουμε κι εμείς, έτσι. Δεύτερον, η σχέση αυτή της μεταφοράς των κονδυλίων στα κράτη-μέλη μπορεί να είναι κίνητρο για τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν τους επιτόπιους ελέγχους γιατί η απειλή θα πρέπει να είναι πως εάν δεν βρείτε το λάθος αλλά το βρουν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε τελείως, ε, σας παίρνουμε τα λεφτά και επίσης θα μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε επικοδομητικά, δηλαδή να πούμε πως εκεί όπου έχουμε πιστεί πως ε, λειτουργούν ε, σωστά οι έλεγχοι, δεν θα κάνουμε εμεί παραπάνω ελέγχους γιατί εμπιστευόμαστε το κράτος μέλο. Δηλαδή να αντιστρέψω αυτό το οποίο λέει ο κύριος Πίπερ. Εκεί όπου έχουμε την αίσθηση πω μπορούμε να βασιστούμε στο κράτος μέλο, γιατί έχει αποδειχτεί πως εργάζονται σωστά και διαχειρίζεται σωστά τα λεφτά μπορούμε να μειώσουμε του ελέγχου. και αντιστρόφως βεβαίω. έτσι. Αύξηση των ελέγχων εκεί όπου βλέπουμε πώ. Ε, έχουμε φοβερά ποσοστά ασφάλματος και έπρεπε να έχουμε περισσότερους ελέγχους. Είναι κοντά σε αυτό το οποίο λέτε, έτσι, δηλαδή να το δούμε ένα χώρα. Νομίζω λοιπόν πως εάν ε, πάμε προς αυτή την κατεύθυνση θα έχουμε κάτι το επικοδομητικό. Ε, επίσης, άλλο ένα ερώτημα προς τον κύριο Επίτροπο, το οποίο προέκυψε από την απάντηση των ερωτήσεων. Στην ερώτηση 53 γάμα μας λέτε πως επί της αρχής αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 6 χώρες οι οποίες δεν έχουν επιφυλάξεις ε, για το θέμα των ιδίων πόρων με βάση τον ΦΠΑ. Ποιες είναι αυτές οι χώρες? θα ήθελα να μας πείτε. Όλοι είμαστε ε, υπέρ του να κατονομάζουμε εδώ πέρα τις ε, χώρες. Οπότε, καλό είναι νομίζω να προσπαθήσουμε να δούμε τι γίνεται με, τα, με τους ίδιους Αλλά το σημαντικό ερώτημα είναι μετά τι συμπεράσματα βγάζουμε για τα άλλα κράτη-μέλη. Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτά τα έξι κράτη-μέλη και για τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ, Γιάν Μιλντερ. Uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς το ελεκτικό συνέδριο καταρχάς, αλλά θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτήν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα υψηλότερο ποσοστό σφάλματος γιατί χρησιμοποιείται ένας άλλος τρόπος υπολογισμού του σφάλματος. Ξέρετε ότι ε, ενδεχομένως να μην δικαιολογείται να χρησιμοποιούμε το σύστημα αυτό για όλα αυτά τα χρόνια, ενδεχομένως να πρέπει να τροποποιηθεί το σύστημα υπολογισμού του σφάλματος. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη, δημοσιονομικές διορθώσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Και όλα αυτά τα έτη που έχουν παρέλθει έχουμε πει ότι το ποσοστό σφάλματος είναι υψηλότερο, αλλά το λεκτικό συνέδριο είχε λάβει υπόψη του τις δημοσιονομικές διορθώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, τότε λέγεται ότι το ποσοστό σφάλματος θα ήταν χαμηλότερο. Αυτό εμένα μου ακούγεται εξ αρχής λογικό. Αν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους εντοπιστεί σφάλμα και διορθωθεί και ληφθεί υπόψη, τότε προφανώς κατεβαίνει και το ποσοστό του σφάλματος. Και αν δεν κάνω λάθος, άλλη άποψη έχει το λεπτικό συνέδριο, γιατί μας ζητά να ακολουθήσουμε κάποιους διεθνείς κανόνες. Μπορεί να αναφερθεί λίγο περισσότερο σε αυτό το λεκτικό συνέδριο. Τελευταία τώρα παρατήρηση να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι έχει καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες προκειμένου να συνεργάζονται καλύτερα οι εθνικές αρχές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις δηλώσεις κάλυψης δαπανών. Ευχαριστούμε επίση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι προσπάθειε που έχει καταβάλει όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα και το σύστημα των management declarations, μια καινοτομία στο καινούριο αυτό σύστημα, δηλαδή δηλώσει διαχείριση. Θα υπάρχει ένα ομοιόμορφο μορφότυπο για τι δηλώσει αυτέ σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Ανδρέασεν. Εκτός μικροφώνου. The is not ε, There is a lot of Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε διάφορες απόψεις για τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος, καθώς επίσης και τις ενδεχόμενε συνέπειες στις δημοσιονομικές διορθώσεις. Από ό,τι κατάλαβα, οι δημοσιονομικές διορθώσεις αποτελούν πλέον την μαγική λύση για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την χρήση και την δαπάνη των κοινοτικών κονδυλίων. Θα ήθελα μία αποσαφήνιση από εσά και από το ελεκτικό συνέδριο, κύριε Επίτροπε, γιατί από ό,τι φαίνεται είπατε ότι το 2012 οι δημοσιονομικές διορθώσεις δεν προσαρμόστηκαν προκειμένου να υπολογιστεί το ποσοστό σφάλματος για το έτος αυτό και η εκπρόσωπος του Ελεκτικού Συνεδρίου μας είπε ότι έγινε όμως κάτι τέτοιο και ότι αφαιρέθηκαν τελικά δημοσιονομικές διορθώσεις, συλλήφθηκαν υπόψη στον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος. Μία άλλη ερώτηση. Όσον αφορά τις ε, δηλώσεις αυτές ε, δαπανών, πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι ε, αντιμετωπίζουμε με απόλυτη τιμιότητα τους Ευρωπαίους φορολογούμενους κάθε φορά που λέμε ότι Όντως, όταν εντοπίσαμε ένα σφάλμα στις δηλώσεις ε, δαπανών των κρατών μελών, ζητήσαμε όντως από το κράτος αυτό να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές και διορθώσεις και ουσιαστικά δεν καταβάλαμε χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να λάβει το κράτος αυτός. Το, αυτό με συγχωρείτε. Όσον αφορά τώρα τις δημοσιονομικές διορθώσεις, σίγουρα συμφωνώ με αυτά που είπατε, αλλά πολύ συχνά έχουμε πληρωμές που γίνονται σε επιμέρους οργανισμούς και υπηρεσίες και όχι μόνο στην κεντρική κυβέρνηση. Οι καθαρές ή κατά αποκοπήν δημοσιονομικές διορθώσεις όμως είναι κάτι το οποίο απαιτείται ή γίνεται σε σχέση με την κεντρική μόνο κυβέρνηση. Αν τα χρήματα αυτά δεν συλλέγονται τελικά από τον τελικό δικαιούχο, τότε ουσιαστικά ο, Ευρωπαϊκός, ο Ευρωπαίος φορολογούμενος είναι αυτός ο οποίος συμβάλλει με επιπρόσθετα χρήματα, με επιπρόσθετα κονδύλια για να καλύψει τις νέες δαπάνες που προκύπτουν. Θεωρώ εδώ πέρα ότι δεν έχουμε σωστή προληπτική προσέγγιση όσον αφορά την κακή διαχείριση και χρήση των ε, κοινοτικών κονδυλίων. Ως προς αυτό λοιπόν, ποια προληπτικά μέτρα μπορείτε εσείς να προτείνετε προκειμένου να μην έχουμε κακή διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ορτής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μέλη του, του συνεδρίου. Θέλω κάτι να διευκρινίσουμε, γι' αυτό και σας ερωτώ από ό,τι κατάλαβα αυτή η επιτροπή που ο συγκεκριτής κύριος που υπηρεπίθεν στον κύριο Μπαρόσο αφορά μια αλλαγή στη διαδικασία όσον αφορά τις δημοσιονομικές καθαρές διορθώσεις. Ισχύει αυτό ή δεν κατάλαβα καλά. Πότε θα τεθεί σε ισχύ και ποια θα είναι ακριβώς η νέα διαδικασία που θα επιφέρει την αλλαγή. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Τσίγματα Μπαλτσίτης, παρακαλώ. E, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, έχω και εγώ μια συντομή ερώτηση. Μια που επί σειρά ετών συζητούμε το πώς θα θεσπιστεί ένα νέο σύστημα, μια νέα μέθοδος, ε, όμως ε, διαπιστώνουμε ότι και σήμερα έχουμε ε, πάρα πολλές αδυναμίες στην μέθοδο που εφαρμόζουμε. Εσείς δεν συμφωνείτε ότι χρήσιμο θα ήταν να καταλήξουμε στο ότι επίκεντρο της προσοχής μας θα πρέπει να είναι το ποσοστό σφάλματος όμως, επίσης, θα πρέπει να προσέξουμε και τις ανακτήσεις από τα κράτη-μέλη προς τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Και έτσι να έχουμε ένα διτό, διπλό σύστημα ελέγχου και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει τώρα κάποιος άλλος τον λόγο. Κοιτάω και την ώρα. Είμαστε ακόμα εντός της ώρας που έχουμε προβλέψει, αλλά πρέπει να βιαστούμε λίγο για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να απαντήσετε κύριε Σέμετα και μετά θα δώσω τον λόγο και στο ελεγκτικό συνέδριο. Κύριε Επιτροπέ. Θα προσπαθήσω, λέει ο κύριο Σέμετα, να απαντήσω με κάποιο συστηματικό τρόπο, γιατί πολλές ερωτήσεις μοιάζουν μεταξύ τους. Οπότε πρώτα-πρώτα, να δούμε το ζήτημα των διορθώσεων και των ανακτήσεων, όπως ε, αναφέρθηκε από τον εισηγητή, τον κύριο Πίπερ και από την κυρία Αντρέσεν. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να είμαστε σαφέστατοι δεν ζητούμε από το ελληνικό συνέδριο να ε, καλύψει με τις καθαρές διορθώσεις το ποσοστό ασφάλμα των, των συγκεκριμένων χρήσεων. Όμως, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η έλεγχη από πλευρά Επιτροπή έχουν πολιετή χαρακτήρα. Άρα δεν ε, έχουν στόχο συγκεκριμένη χρήση. Αλλά υπάρχει μια σειρά ελέγχων. Ξεκινούμε από κάποιες προληπτικές δράσεις όπως ε, διακοπές, αναστολές πληρωμών σε πτώση που τα κράτη-μέλη δεν ε, εφαρμόζουν με το σωστό τρόπο το σύστημα Κατόπιν έχουμε τις ε, δημοσιονομικές διορθώσεις και τις ανακτήσεις που είναι τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των ελέγχων. Και έτσι εξηγείται γιατί θεωρούμε ότι χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αυτός ο πολιετής χαρακτήρας των ελέγχων μας. Και ο κύριος Πίπερ ότι έχουμε το 2012 οπότε ε, διορθώσεις συνδέονται με τις χρήσεις του 2006. Ναι, είναι αλήθεια ότι πολλές από αυτές τις διορθώσεις έγιναν επί του προπολογισμού των ετων 2000-2006. Αυτό όμως σημαίνει ότι το σύστημα αποδίδει και είναι πάρα πολύ πιθανό τα ασφάλματα τα οποία διεπράχθησαν το 2012 πρόκειται να διορθωθούν εις το μέλλον λόγω του πολιετούς χαρακτήρα των ελέγχων. Γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται αυτό το χαρακτηριστικό των ελέγχων να ληφθεί υπόψη. Και ήδη το Ελληνικό Συνέδριο κινήθηκε προς αυτήν την ε, πολιτική μεθοδολογία. Δεν ασκεί ελέγχου στις ε, πρώιμες πληρωμές αλλά και έλεγχο στην εκαθάριση αυτών των πρώιμων πληρωμών. Ε, ε, γίνεται αυτή η προπληρωμή και μια χρήση και η καθάριση την επομένη χρήση ή σε κάποιες φάσεις, ε, σε κάποιες περιπτώσεις της άμεσης διαχείρισης όπου έχουμε κάποιες εξωτερικές πολιτικές οπότε η καθάριση των προπληρωμών γίνεται ε, σε καποιες φασεις σε καποιες περιπτωσεις της αμεσης διαχειρισης οπου εχουμε καποιες εξωτερικες πολιτικες οποτε η εκαθαριση των προπληρωμων γινεται σε υστερη φάση των πληρωμών. Πάντως αυτό το οποίο εμείς ε, λέμε, αυτό το οποίο ζητούμε, είναι αυτό να κάνετε, αυτό να λάβετε υπόψη. Κύριε Ανδρέας, αν ε, ρωτήσατε συγκεκριμένα τι έλαβε υπόψη το ελληνικό συνέδριο και τι δεν έλαβε. Ε, ας απαντήσει καλύτερα το ελληνικό συνέδριο. Πάντως το θέμα είναι ότι το ελληνικό συνέδριο λαμβάνει υπόψη τις διορθώσεις οι οποίες έγιναν τη συγκεκριμένη χρήση του ελέγχου και τη διόρθωση όσον αφορά τον τελικό δικαιούχο. Οπότε, έτσι, γίνεται όσον αφορά τις πληρωμένες και λαμβάνονται υπόψη αυτές οι διορθώσεις Αυτό δεν είναι σε μεγάλη μεγέθου. Πάντως πρέπει να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση. Μπορεί να πάρει τα χρήματα από τους τελικούς ε, δικαιούχους. Τα κράτη-μέλη το κάνουν αυτό. Ο δικός μας ρόλος είναι να προστατεύσουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση με τι διορθώσει. Και τα κράτη-μέλη μπορούν να ανακτήσουν τα χρήματα από τον τελικό δικαιούχο. Και έτσι προστατεύουν τον εθνικό προπολογισμό. Αν όμως αποφασίσει το κράτος μέλος, θεωρήσει ότι επέτευθαν οι στόχοι κάποιου προγράμματος και δεν χρειάζεται να ανακτηθούν χρήματα από τον τελικό δικαιούχο, τότε πρόκειται για απόφαση των πολιτικών αρχών του κράτους μέλους. Να μην ανακτήσουν τα χρήματα από τον ε, δικαιούχο και να τον χρηματοδοτήσουν τον δικό προπολογισμό. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η προστασία του προπολογισμού της Ένωσης. Έτσι λοιπόν εργαζόμαστε εντατικά και προσπαθούμε να αυξήσουμε τις διορθώσεις και τις ανακτήσεις. Από πλευρά τη Επιτροπής το θέμα τώρα είναι το ότι κατόπιν των διορθώσεων τα κρατή-μέλη θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα προγράμματα που είναι στραβά με κάποια καινούργια. Κάτι το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. το έχετε εγκρίνει εσείς και το Συμβούλιο και εμείς ως φύλακες των συνθήκων. Επομένως θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις αυτές όπως θεσπίστηκαν από τους συνομοθέτες. Αυτά τα λίγα λόγια όσον το σύστημα των διορθώσεων και ανακτήσεων. Και τώρα, για να δούμε τι γίνεται με την καθαρή διόρθωση πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Πίπερ για τις ε, παρατηρήσεις του για το πώς αυτές οι διορθώσεις θα ενταχθούν στο σύστημα της πολιτικής συνοχής. Από οπτικής γωνίας πολιτικής θα πρέπει να σα τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο, όσο γίνεται περισσότερο. Όσο επιτρέπει η νομοθεσία. Οι συνομοθέτες ξεκαθάρισαν και όρισαν ποιος είναι ο ορισμός σοβαρής αδυναμίας, του δημοσιονομικής διόρθωσης. Προσπαθήσαμε δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Όσο με τους ορισμούς αυτούς, αλλά δεν πάμε παραπέρα να ξεπεράσουμε αυτούς τους ορισμούς οι οποίοι έχουν θεσπιστεί νομοθετικά. Τώρα επομένως Βλέπουμε τι γίνεται με την κατοξιδότηση πράξη σε, επίπεδο υπηρεσιών. Να συνοηθούμε ούτως ώστε να δούμε πώς θα εκφραστούν και οι δικές σας απόψεις. Πάντως, συμφωνώ με την απόψή σας, ότι δηλαδή θα πρέπει αυτή η διαδικασία να γίνει όσο πιο αυτόματα είναι δυνατόν. Αλλά θα πρέπει να τηρήσουμε τους ισχύοντες κανόνες. Φερρυπίν ορίζει νομοθεσία ξεκάθαρα ότι όταν έχουμε έλεγχο κατά διάρκεια του οικονομικού έτους δεν μπορούμε να επιβάλλουμε καθαρή διόρθωση. Όμως μπορούμε να την ασκήσουμε αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 φορές του επομένου έτους όλα όσα πρέπει να υποβληθούν τα κρατημέλη, οπότε έγινε ο έλεγχος δηλαδή και έχει διαπιστωθεί ότι κάτι πάει στραβά σε αυτό το κράτος μέλος. Υπάρχουν κάποια σφάλματα. Τότε μόνο μπορούμε να έχουμε αυτή την καθαρή διόρθωση. Αυτά προβλέπει η νομοθεσία. Εγώ και οι συνάδελφοι έχουμε την αρμοδιότητα αυτή και στην κατεξοδοτική πράξη ορίσαμε τι είναι η καθαρή διόρθωση. Δώσαμε τον ορισμό, αλλά δεν μπορούμε στην κατευθυντική πράξη να πάμε αντίθετα προς όσα ορίζει η νομοθεσία. Τώρα είμαστε σε επίπεδο διαβούλευση των υπηρεσιών μας για αυτή την εξουσιακή πράξη. Πρόκειται να εγκριθεί τον Φεβρουάριο μέσα σε ένα μήνα. Όσον αφορά τώρα Τι ερωτήσει για την Όλαφ από τη κυρία Γκρέσλε. Πρώτα πρώτα. Θα πρέπει να είμαι σαφής. Το στις απαντήσεις. Ότι η Όλαφ ουδέποτε κατέγραψε συνομιλίες ε, ιδιωτών. Κατ' εξαίρεση σε μια περίπτωση η Όλαφ συνεργάστηκε. με τέτοια καταγραφή συνομιλιών. Αλλά σύμφωνα με τους νομικούς μας συμβούλους η εν λόγω ενέργεια προβλέπεται από την νομοθεσία που διέπει την όλα. Και αυτό το ετυπώνουμε ξεκάθαρα στην έγγραφη απάντηση προς την ερώτησή σας. να τον τώρα να δούμε τα πιο πολιτικά στοιχεία του θέματος κυρία Κυριασλέα. Γνωρίζετε ότι πέρσι είχαμε αυτή την πρόταση για τον EPPO και διατυπώσαμε την πρόταση για κάποιες ε, άλλες ιδέες, για κάποιες διαδικαστικές εγγυήσεις για τα φυσικά πρόσωπα. Τώρα δε επεξεργαζόμαστε τι επιλογές υπάρχουν όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις για την Ιωνή νομική έγκριση των διατάξεων που τα θεσμικά όργανα και πιστεύω ότι με αυτή την πρόταση που θα έχει διατυπωθεί οριστικά τον Μάρτιο. Θα κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και θα εξασφαλίσουμε περαιτέρω τις διαδικαστικές ή δικονομικές εγγύσεις για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή στην έρευνα. Τώρα, όσον αφορά την αναθεώρηση για το προσωπικό. Ήταν θετικό το ότι ενήργησε σχετικά η Όλαφ, ε, το, το, προσωπικό ε, αντέδρασε, αποκρίθηκε τέλο πάντων όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και αυτή η μεταρρύθμιση θα χρησιμοποιηθεί όσον αφορά την πρώτη ε, Παρασκευή, την προετοιμασία μιας νέας στρατηγικής από πλευράς Όλαφ και έχουμε τις συγκεκριμένες απαντήσεις, συγκεκριμένες ερωτήσεις για την Όλαφ. Και πιστεύω ότι αυτά τα στοιχεία πρόκειται να εξυπηρετήσουν το πώς θα έχουμε μια συνολική, πλήρη στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους. και επομένως θα υπάρξει τέτοιος διάλογος για να μπορέσουμε να δούμε την αίσθηση για τους ανθρώπινους πόρους, να την ολοκληρώσουμε, να την προετοιμάσουμε και να την εφαρμόσουμε στη συνέχεια. Οπότε, σε σχέση με την κύριο Γκάια, για τους ίδιους πόρους. Δεν θυμάμαι ακριβώς για ποια κράτη-μέλη μας μίλησε, οπότε καλύτερα εγγράφως να συνοηθούμε και να του δώσουμε τα στοιχεία αυτά που θέλει για τα κράτη-μέλη με τις επιφυλάξεις. Στην, έγραφη, απάντηση, στην απάντηση μάλλον για την διόρθωση νομίζω έμεσα κάλυψα και την ερώτηση του κυρίου Μίλτερ όσον αφορά το τι κάνουμε με το ποσοστό σφάλματος. Την διαχείριση, τον μορφότυπο της, διαχ... της δήλωσης διαχείρισης. Μιλάμε για δύο εβδομάδες το πολύ. Οπότε και θα παρουσιάσουμε αυτόν τον μορφότυπο ή στην ομάδα εργασίας που ασχολείται με την εθνική αυτή δήλωση. Νομίζω κάλυψα και τα όσα είπε ο κύριος Μπαλτσίτης και η κυρία Βιλέλια. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, ευχαριστώ να τις απαντήσω και εκείνες. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, καθαρίσατε πως ε, η Κομισιόν βασίζεται σε κάποια νομική βάση όσον αφορά τις ε, δημοσιονομικές διορθώσεις. Απλά να πω πως για την Επιτροπή μας έχει μεγάλη σημασία να αλλάξει η συμπεριφορά των δικαιούχων. Εάν τα κράτη-μέλη πληρώνουν τα χρήματα για λογαριασμό των δικαιούχων που έκαναν κατάξη των κονδυλίων, δεν αλλάζει η συμπεριφορά τους. Οπότε εμείς ως Επιτροπή ελέγχου του περιπολογισμού επιμένουμε να επιβληθούν κυρώσεις σε όσους ε, ε, έκαναν κακή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εσείς ε, βεβαίως βασίζεστε στην νομοθεσία, ίσως μπορούμε να σας ενθαρρύνουμε να αλλάξετε την νομοθεσία, να μιλήσετε με τα κράτη-μέλη. Τώρα δεν θέλω να ανοίξουμε ένα δεύτερο γύρο συζητήσεων, αλλά αν υπάρχουν ερωτήσεις να σας υπενθυμίσω και το χρόνο και να δώσω τώρα το λόγο στο ελεκτικό συνέδριο. η κυρία Γκρέσλε. Α, ναι. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, αλλά έθεσα τρεις ερωτήσεις και απαντήθηκαν οι δύο, ή τέλος πάντων κάπως απαντήθηκαν. Η τρίτη ερώτηση τώρα, γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος μέχρι ο Βέλγος δικαστής, ο κύριος Φαν Έσπεν, να μπορέσει να καλέσει σε απολογία τους τρεις ανθρώπους του Όλαφ. Δηλαδή πέρασε ένας χρόνος σχεδόν. Γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος. Δεν είναι δυνατόν. Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρειάστηκε έξι μήνες για να διαβιβάσει την πρόσκληση του κυρίου Φανέσπεν και σε τρεις βουλευτές, μεταξύ των οποίων και σε εμένα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα έναν Βέλγο ανακριτή, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του και μια συνολική αδιαφορία των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν για την έρευνα του προσωπικού που κάνατε, αλλά υπάρχουν δύο έρευνες του προσωπικού. Εγώ θα ήθελα να μας δώσετε και την δεύτερη έρευνα που αφορά που έγινε από την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, όχι αυτή που έκανε ο, Όλαφ. Βεβαίως εννοείται αμνησία, έτσι, και όχι ανάμνηση, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Ναι, Πράγματι, δεν χρειάστηκε ένας χρόνος. Έξι μήνες χρειάστηκαν όντω για να απαντηθεί το ζήτημα αυτό. Ήταν ε, δυστυχώ ένα διοικητικό λάθος στην επεξεργασία των εγγράφων ε, εντός του Όλαφ και σύμφωνα με τις ε, πληροφορίες μου γιατί ενημερώνομαι τακτικά από τον Όλαφ αυτή τη στιγμή συνεργάζονται πλήρως με τις δικαστικές αρχές που διερευνούν τις ε, περιπτώσεις, τη λεγόμενη περίπτωση Νταλίκ. Και δεν έχουμε παράπονα ή οχλήσεις ε, από τις δικαστικές αρχές ε, για αυτό το ζήτημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν που αναφέρεται ήταν μια, ένα τυχές διοικητικό λάθος στην επεξεργασία των εγγράφων. Μάλιστα. Τώρα με, με το θέμα του κοινοβουλίου ξέρετε πως υπάρχουν και συμπτώσεις. Λοιπόν, τον λόγο τώρα έχει το ελεγκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω πρώτα στον κύριο Μούλτερ. Δεν αλλάξαμε τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού σφάλματος. Απλώς δεν χρησιμοποίησαμε κάποια ποσά προκαταβολών. Το υφιστάμενο σύστημα μας επιτρέπει να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για τις άμεσες πληρωμές και δεν έχουμε ακόμα εναρμονισμένη προσέγγιση. Ξέρετε ότι ε, αν δεν ήμασταν σε θέση να έχουμε κάποια στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουδέποτε θα είχαμε καταφέρει να καταλήξουμε σε κάποια εναρμόνιση. Ευχαριστούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, ε, μπορούμε να αναφερθούμε και στο μέλλον σε κάποια νέα στοιχεία τα οποία θα ισχύσουν για τον τομέα της συνοχής. Ο κύριος Πίπερ, η κυρία Σένα, ο κύριος Μούλτερ αναφέρθηκαν στο ότι το ποσοστό σφάλματος θα είχε ευθυγραμμιστεί με αυτό το περσινό αν είχαμε λάβει υπόψη μας τις καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις. Ως προς αυτό να σας πω ότι προσπαθήσαμε να καταλάβουμε το επιχείρημα αυτό, ωστόσο δεν έχουμε καταφέρει να καταλάβουμε ακριβώς πώς υπολογίζεται αυτό το ποσοστό σφάλματος ακόμα και αν είχαμε λάβει υπόψη μας τις δημοσιονομικές διορθώσεις του 2012. Θα καταλήγαμε ουσιαστικά πάλι στο ίδιο ποσοστό. 4,5%. Μείον 3,9%. Βρισκόμαστε σε ποσοστό 0,8 όσον αφορά τη διαφορά. Τώρα, τι λαμβάνουμε υπόψη και τι όχι στο συνέδριο. Λέγεται ότι μόνο λαμβάνουμε υπόψη μας το ζήτημα της αντικατάστασης σε επίπεδο προγράμματος. Όντως αυτό λαμβάνεται υπόψη και το βλέπετε αυτό στο κεφάλαιο 1, σε ένα παράδειγμα το οποίο δίνει το συνέδριο για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ήδη όμως στο παρελθόν όταν ένα κράτος μέλος είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε κάνει εσφαλμένη δήλωση δαπανών, θα είχε τότε ακόμα το δικαίωμα να αποσύρει την δήλωση αυτή και να αποσυρθεί η δήλωση, βέβαια το συνέδριο δεν πρόκειται να έρθει και να πει ότι θα πρέπει να αντικαταστήσετε συγκεκριμένε δαπάνε στο έργο αυτό. Οι αποσυρώμενε δαπάνε ουσιαστικά αφαιρούνται αυτόματα και από το ποσοστό σφάλματο. Γιατί ουσιαστικά δεν εξετάζουμε ποτέ, το λαμβάνουμε υπόψη μα τη δήλωση δαπάνη η οποία τελικά δεν ελήφθη υπόψη. Έχει να κάνει δηλαδή με εσφαλμένο πρόγραμμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη πρέπει να υποβάλουν μια νέα δήλωση κόστους προκειμένου να έχουμε ξεκάθαρες δηλώσεις δαπανών οι οποίες θα ενταχθούν στην τελική δήλωση αφού του κράτους μέλους. Σε πολλές περιπτώσεις δεν λαμβάνουμε υπόψη, όπως σας είπα, τις εσφαλμένες αυτές δηλώσεις, οι οποίες σε κάποιο στάδιο αποσύρονται από το κράτος μέλος. Λέμε επίσης ότι θα πρέπει οι δαπάνες να καταβάλλονται με τρόπο νόμιμο και κανονικό. Στην αντίθετη περίπτωση έχουμε κάποιες αρνητικές συνέπειες για τον κοινωνικό προπολογισμό. Για το 2013 είδαμε ανακτήσεις, ενώ το 2012 είχαμε μόνο καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι προστατεύεται ο κοινοτικό προπολογισμό και ότι αυτό ουσιαστικά μόνο κοιτάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν όμω γίνει κάτι τέτοιο, τότε δεν θα καταφέρουμε να έχουμε συμπεριφορά, αλλαγή συμπεριφορά των κρατών μελών. Εμεί με τη δική μα τη στάση έχουμε επιφέρει μια αλλαγή στη στάση των κρατών μελών. Ο κύριο Σεμέτ επίση μα είπε ότι στην υφιστάμενη περίοδο προγραμματισμού οι διακοπές, αναστολές πληρωμών είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο που έχουμε προκειμένου να πείσουμε τα κράτη-μέλη να δαπανούν σωστά τα κοινοτικά κονδύλια. Και σίγουρα δεχομένω θα είναι το πιο ισχυρό μέσο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή και εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή. Σας υποσχέθηκα ότι ε, θα αναφερθώ και σε κάποια θεωρητικά ζητήματα μαζί σας όσον αφορά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, γιατί ο κύριος Μούλτερ έθεσε ανάλογο ερώτημα και θα αναφερθώ όντω στην ε, προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία τα κράτη-μέλη πρέπει να ανακαλύψουν και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Ο κύριος Πίπερ μας έδωσε κάποια παραδείγματα και μας έδωσε και κάποιες εξηγήσεις για το πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό. Πρέπει να σας πω όμως ότι το λεκτικό συνέδριο όντω κάνει ελέγχους στο τέλος του έτους, άρα στις 15 Φεβρουαρίου έχει ήδη ολοκληρώσει τον βασικό του έλεγχο για το έτος αυτό το προηγούμενο δηλαδή, το ελεκτικό συνέδριο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλα τα σφάλματα τα οποία έχουμε εντοπίσει μπορούν πλέον να διορθωθούν από τα κράτη-μέλη, έχουν γνωστοποιηθεί στα κράτη-μέλη. Εμείς δεν λέμε ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσετε το έργο του ελεκτικού συνεδρίου για να διορθώστε τα σφάλματά σας. Το πρόβλημα είναι ότι όταν βρισκόμαστε στο έτος νη συνένα, δεν μπορούμε να κάνουμε εμεί τον ίδιο αυστηρό έλεγχο με αυτό που κάνουμε για το έτος εκείνο το οικονομικό το οποίο είχε ολοκληρωθεί. Δηλαδή, στην φάση νη συνένα δεν είμαστε σε θέση να έχουμε σφαιρική εικόνα του ποσοστού σφάλματος. Το ελεκτικό συνέδριο ουσιαστικά βασίζεται στα όσα λέει η συνθήκη και ολοκληρώνει πάντα τον έλεγχό του αφού ολοκληρωθεί το οικονομικό έτος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε από κοινού πώς μπορεί ενδεχομένως να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου και να γίνουν κάποιες προσαρμογές για τα μελλοντικά έτη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Καλουλάιντ, ο κύριος Πίπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη βοήθειά τους, για τις προτάσεις τους, τη συμβολή τους. Θα ήθελα να αναφέρω δύο την ακόμη. Μας ε, προβληματίζουν τα παραθυράκια που υπάρχουν όσον αφορά το σύστημα των διορθώσεων. Ας πούμε, πώς θα δώσουμε τον ορισμό της ε, σημαντικής παραβάσεως. Θα πρέπει να βρούμε κάποιον ευέλικτο ορισμό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει διάθεση να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά τους κοινωτικούς πόρους. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν στεγανές, όπως είπαν οι σχετικές διατάξεις. Δεν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαλαρώσει τον έλεγχο της επί των κρατών μέλων. Το αντίθετο. Να υπάρχει η άμεση δειγματοληψία. πέραν των οικονομικών ελέγχων. Και αυτό να γίνεται με τρόπο αυτόματο και αυτοδίκαιο για τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν εμφανίσει κάποιε αδυναμίε, κάποια προβλήματα στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Επίτροπο και δίνει το λόγο. Ε, μάλλον, συγγνώμη, ευχαριστεί, ευχαριστεί τον Επίτροπο που ήρθατε, που συζητήσαμε, λέει. Και Θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή. Διαπιστώσατε ότι κάποιοι βουλευτέ δεν ικανοποιήθηκαν 100% με κάποιε απαντήσεις, οπότε παρακαλώ σκεφτείτε τις ερωτήσεις. Ε, μπορείτε να παράσχετε περαιτέρω ενημέρωση. Πάντως σα ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα το πρωί εδώ για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Σα ευχαριστούμε.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πολλά σημεία στη μερίσια διάταξη. Σας περάσουμε αμέσω στο επόμενο σημείο λοιπόν. Σημείο παριθμών 9 σε δύο τμήματα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Κάθριν Ντέι, Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας καλωσορίζουμε κυρία Ντέι. Ας συζητήσουμε πρώτα τα ζητήματα που άπτονται της απαλλαγής από κοινού και στη συνέχεια θα περάσουμε στο ζήτημα των ερευνών της Όλαφ. Όσον αφορά λοιπόν την απαλλαγή 2012, θα ήθελα να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου, τον κύριο Ντομέ Μουγκουρούζα, και του δίνω ευθύ αμέσω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, αξιότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κεφάλαιο υπαριθμών 9 της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται στις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ στο κεφάλαιο 9 αναφερόμαστε σε όλα τα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε και κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις και συστάσεις που αφορούν επιμέρους όργανα και θεσμικά και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστοιχούν ουσιαστικά στο 7% των συνολικών πληρωμών που γίναν το 2012, οι διοικητικές δηλαδή δαπάνες και οι μισθοί, επιδόματα, συντάξεις συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες αυτές, καθώς επίσης και δαπάνες που έχουν να κάνουν με τα κτίρια, τις υποδομές πληροφορικής κτλ. Το 2012 το Ελεκτικό Συνέδριο έχει επιφέρει τρεις βασικές βελτιώσεις όσον αφορά το σχετικό έλεγχο που γίνεται για τις διοικητικές δαπάνες. Η πρώτη βελτίωση έχει να κάνει με τον αριθμό των ελέγχων όσον αφορά συγκεκριμένε συναλλαγές που έλαβαν χώρα. Το 2012 το ελεκτικό συνέδριο έκανε διάφορους αντιπροσωπευτικούς ελέγχους 151 συνολικά συναλλαγές ε, ελέγχθηκαν, ενώ στο, το 2012 είχαμε 56 τέτοιες συναλλαγές οι οποίες έτυχαν ελέγχου. Καταλαβαίνετε ότι μέσω της αύξησης των ελέγχων αυτών των συναλλαγών καταφέρνουμε να έχουμε μια πιο δικημενική εικόνα όσον αφορά την οικονομική κατάσταση. Δεύτερη βελτίωση, καταφέρνουμε να βελτιώσουμε κάποια λάθη τα οποία γίνονται στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών. Το 2012 είχαν εντοπιστεί σημαντικά σφάλματα όσον αφορά τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και των προμηθειών που συνέβαλαν πάρα πολύ στην αύξηση του ποσοστού σφάλματος. Μέσω των βελτιώσεων που καταφέραμε να επιφέρουμε το 2012 έχουμε πλέον ένα βελτιωμένο σύστημα επιθεώρησης όσον αφορά τις εν λόγω αυτές συναλλαγές. Ως προς αυτό το ελεκτικό συνέδριο κάνει πλέον ενδαλεχείς επιθεωρήσεις δύο θεσμικών οργάνων που ε, επιλέγει κάθε έτος. Το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήταν τα δύο αυτά θεσμικά όργανα τα οποία είχαν ελέγχου. Το 2013 θα συνεχιστεί ο έλεγχος αυτός και θα καλύψει τις ε, σχετικές συναλλαγές προμηθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά αυτόν τον τρόπο το ελεγκτικό συνέδριο θα είναι σε θέση του χρόνου να έχει μια πιο σφαιρική εικόνα στην έκθεσή του για τις αδυναμίες και τα προβλήματα τα οποία είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών. Όσον αφορά τώρα τα συμπεράσματά μας, όπως και τα προηγούμενα έτη, έτσι και φέτος, το πόρισμά μας είναι θετικό και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι συναλλαγές που έχουν να κάνουν με τις διοικητικές δαπάνες το 2012 ήταν από ουσιαστική πλευρά νόμιμες και κανονικές. Πιο συγκεκριμένα τώρα, το λεκτικό συνέδριο εντόπισε ότι στις 151 συναλλαγές που ήλεγξε Μία λοιπόν μόνη είχε σημαντικό σφάλμα. Σε όλε τι υπόλοιπε συναλλαγέ το ποσοστό σφάλματο ήταν μηδενικό. Το ελεκτικό συνέδριο επίση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα επιτήρησης και ελέγχου για τις δυτικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων συνάδουν με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελεκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά το σύστημα επιτήρησης και ελέγχου. Ωστόσο, εντόπισε κάποιες αδυναμίες όσον αφορά τη διαχείριση των κοινωνικών επιδομάτων, όπως και τα προηγούμενα έτη, και βλέπουμε ότι ο βασικός λόγος προκύπτουν οι δυναμίες αυτές είναι η έλλειψη συγκεκριμένων πληροφοριών για τα κοινωνικά αυτά επιδόματα και τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν πολλές φορές μέλη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό όμως επίπεδο, περισσότερο τα αποσπασμένα λοιπόν μέλη. Έχουν γίνει συζητήσεις ε, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεκτικού Συνεδρίου και θεωρούμε ότι θα πρέπει πλέον από τις υπηρεσίες πληρωμών των επιδομάτων αυτών και των αποζημιώσεων να αρχίσει να χρησιμοποιείται ένα νέο, πιο αυστηρό σύστημα. Εκ του σύνεγγυ πρόκειται στο μέλλον να παρακολουθήσει το νέο αυτό σύστημα το λεκτικό συνέδριο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είμαι στην πλήρη διαθεσή σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις ή αποσαφηνήσεις που θέλετε να ζητήσετε από μένα. Σας ευχαριστώ επίσης για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ, κύριε Τόμε Μουγκουρούτσα. Επομένως, τώρα μπορούμε να δούμε τη σκητάλη ή τον εισηγητή. Όχι, μετά. Θα δούμε το λόγο στην κυρία Ντέι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τέτοιου είδους θετική γνωμοδότηση από πλευρά του συνεδρίου. Ευχαριστώ που με καλέσατε για σήμερα το πρωί εδώ για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της ετησίας εκθέσεως του συνεδρίου του 2012. Έχω έτσι την ευκαιρία σύντομα να σας πω δύο λόγια για τα όσα κάναμε που σας ενδιαφέρουν, που είναι αρμοδιότητά σας και βέβαια να συζητήσουμε γενικότερα για αυτά που σας ενδιαφέρουν σήμερα το πρωί. Εγκρίνετε την έκθεση του Προέδρου σας. Πάρα πολύ θετικά τα όσα συμπεράνονται και προσπαθούμε επομένω να βελτιωθούμε, να προοδεύσουμε, να κάνουμε το κάθε χρόνο. Για να δούμε τώρα. Να σταθούμε στα θέματα μεθοδολογίας μας πρώτα-πρώτα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε το άρθρο 3.18 Το έχουμε σωματώσει στην μεθοδολογία μας όπως ζητήσατε. Επίσης όπως προσέξατε η έκθεση μας δημοσιοποιήθηκε πολύ νωρίτερα από ότι προηγουμένως όπως ζητήσατε τώρα επί τη βάση των ε, ε εκθέσεων δραστηριότητα το 2013 είπαμε τον Ιούνιο για το τι έγινε και για τη στρατηγική ενόψη του 2020, δώσαμε ιδιαίτερο βάρο που και αυτό σας ενδιαφέρει και τώρα όσον αφορά το πολιτισμικό πλαίσιο, ε, τώρα θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε πώς θα τα πάμε, θα κάτι μέλη να εφαρμόσουν τα νέα προγράμματα και αφού υλοποιηθούν, εφαρμοστούν τα προγράμματα, θα δούμε τις επιδόσεις των μελών, προγραμματισμός, ε, εκθέσεις για τις επιδόσεις. Αυτά επίσης τα υιοθετήσαμε ως μεθοδολογία και κάναμε όσο πιο γρήγορα γίνεται ό,τι μπορέσαμε για να υλοποιήσουμε τις συστάσεις του ελεγχτικού συνεδρίου. Στον αφορά βάση του προγράμματος, όπως εγκριθήκε από Συμβουλίο και Κοινοβούλιο τέλος ε, παρελθόντος έτους, είπαμε, θα καλύψουμε το προγραμματισμό, τις επιπτώσεις των προγραμμάτων, ε, όλα αυτά στις εκθέσεις τις σχετικές, τώρα πιο συγκεκριμένα, όπως σας είπα, ότι θεωρούσαμε θετικά τα όσα είπε το ελληνικό συνέδριο ε, και επίσης ε, θεωρήσαμε πάρα πολύ θετικά αυτά το οποίο είπε το ελληνικό συνέδριο και επίσης ε, θεωρήσαμε ότι οι έκτακτες εκθέσεις είναι πολύτιμες ε, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε κατά τις πολιτικές μας όλους τους τομείς και βέβαια συμφωνούμε ότι το σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να μετρά τα επιτεύγματα σε σχέση με τις δαπάνες και στην έκθεσή μας προς το Κοινοβούλιο και ιδίως στην τελευταία μας έκθεση θίγουμε αυτές τις πρωτοβουλίες για τις επιδόσεις μας με τη διαχείριση. Τώρα για να δούμε στα πλαίσια του πολιτού προγράμματος του MFF είπαμε ε, εξάντε να, να ελέγξουμε τι γίνεται με τους στόχους μας και κατόπιν όλα αυτά να γίνουν σχέδια προγράμματα διαχείρισης για την αξιολόγηση ex post. Και αυτά μπορείτε να τα δείτε ε, στην ετησία έκθεση δραστηριοτήτων, των στις προηγούμενες αξιολογήσεις και την έκθεση του συνεδρίου. Ε, εμείς Ε, προσπαθήσαμε στο MFF 2014-2020 να επιφέρουμε απλουστεύσεις, να καλύψουμε την προσθέμενη αξία από την εκτέλεση του προπολογισμού της Ένωσης και επίσης να γίνει η μελέτη επιπτώσεων ε, όλων αυτών των πολιτικών μας για την Ευρώπη. Επίσης, φεύγουμε κάποιες ειδικέ διατάξεις για υποπτία. Ε, υποβολή εκθέσεων για, την, ε, για τις επιδόσεις μας και είπαμε σε διάλογο με Κοινοβούλιο και Συμβούλιο θα εξετάσουμε το που πήγαμε καλά, που πήγαμε λιγότερο καλά αλλά θεωρούμε ότι υπάρχουν καινούργια στοιχεία που μας βοηθούν για το μέλλον. Αναφέρθηκα στα προγράμματα διαχείρισης στις εκθέσεις των Γενικών Διευθύνσεων. Όλα αυτά τα αναβαθμίσαμε και έχουμε κάποιες ε, βελτιώσεις, ε, τα διοικητικά προγράμματα, τα προγράμματα δραστηριοτήτων, να τα κάνουμε πιο συγκρίσιμα, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους μορφότυπους για τη διαχείριση και στις αιτήσεις εκθέσεις δραστηριότητας. Επίσης έχουμε ε, οργανώσει κάποιες εσωτερικές ε, αναφορές, εκθέσεις ε, αναθεώρησης και όποιος θέλει να τη χρησιμοποιήσει μπορεί να επισημάνει τα σημεία που του χρειάζονται συγκεκριμένα. Επίσης έχουμε κάποιους ε, δείκτες επιδόσεων και έτσι να δούμε πώς και αυτό θα γίνει πιο χρηστικό για όποιον χρειάζεται. Για τις αιτήσεις εκθέσεις καλύπτουμε επομένως τώρα συνεπώς και συνεχώς τις ε, επιδόσεις. Το ελληνικό συνέδριο ε, τα δει με καλό μάτι όλα αυτά, αλλά θα δούμε τα οριστικά αποτελέσματα στο μέλλον και η νομική βάση όπως εγκρίθηκε θα πρέπει με το δευτερογενές κοινωτικό δίκαιο να συνδυαστεί με τα άλλα εργαλεία που έχουμε να χρησιμοποιηθεί και έτσι να έχουμε αποτελέσματα όσον αφορά την προσθέμενη αξία από την εκτέλεση του κοινωνικού προπολογισμού. Εν κατακλείδη να σας πω τι γίνεται όσον αφορά τα της απλούστευσης, σας είπα για το MFF και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει μια ανακοίνωση για την απλούστευση και επίσης από τη μεγάλη σημασία στο πόσο σημαντικό είναι να πριτανεύσει η απλούστευση όχι μόνο σε αυτή την νομοθεσία αλλά και αυτό να είναι ε, κάτι για το οποίο είναι συνυπεύθυνο και τα κρατημέλη. Όλοι μας θα πρέπει να απλουστεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Έχουμε επίση έκθεση για το πώς προχωρήσαμε μέσω της συναπόφασης. Έχουμε επίσης ε, έναν χάρτη επιδόσεων, κατάλογο επιδόσεων για την απλούστευση και είδαμε ότι για κάποια προγράμματα Έχουμε κάποια υπαχθή, τέλο πάντων βαριά, δυσκίνητη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Έχουμε επίσης ε, βυζαντινολογία όσον αφορά το, τις λεπτομέρειες εφαρμοστικές. Διαδικασία επιτροπών σε διάφορα σημεία και ε, επίσης ε, υπάρχει περιθώριο για απλούστευση και ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση του προπολογισμού. Πάντως ε, τώρα για το MFF έχουμε τις προτάσεις, προχωρήσαμε την απλούστευση και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα τρίτο και τελικό πίνακα επιδόσεων να δούμε τι έχει προτείνει η Κομισιόν, τι έχει προτείνει και τι, τι, απέριψε το Κοινοβούλιο και τι ανέκρινε και, γιατί προέτεινε και τι απέρριψε το Συμβούλιο. Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι έχει μόνο ακαδημαϊκή, ιστορική αξία, αλλά θα βοηθήσει όσον αφορά την υλοποίηση του νέου πλαισίου δημοσιονομικού MFF. Οπότε, να δούμε πού αλλού χωρεί. Απλούστευση και να προχωρήσουμε ένα λόγος. Να μην επισέλθω και σε άλλες λεπτομέρειες, γιατί έχετε τόσα να κάνετε, Πρόεδρε και ευχαρίστω να απαντήσω σε για όσα είπα και όσα δεν είπα. Κύριε Αντέ, σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε. Να σα ευχαριστήσω όμω και ως εισηγητής. αυτή την προσέγγιση πλευρά των επιδοσιών μας, κάτι το οποίο θέλουμε να κυριαρχήσει. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους. Ποιος θέλει τον λόγο, ο κύριος Πίπερ και η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα. Σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία έχετε ήδη κάνει όσον αφορά τον έλεγχο των συστημάτων. Είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Ελπίζω πραγματικά και εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω να τα καταφέρετε εδώ πέρα. Κατά κύριο λόγο μιλάμε για τις δαπάνες. Μιλάμε για ευρωπαϊκά λεφτά, χρήματα των προλογούμενων και εδώ πέρα θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια πράγματα. Πρώτον, στην έκθεση σύνθεσης της Κομισιόν του 2012 όπου αναφέρονται τα συνολικά ποσά που περιγράφονται ως ποσά που περιέχουν κάποιον κίνδυνο και μιλάμε για ένα συνολικό ποσό το οποίο είναι μεταξύ 2,6 και 3,4 δισεκατομμυρίων το ελεγκτικό συνέδριο είπε πως η Κομισιόν άρα παραδέχεται πως το ποστό σφάλματος στις δαπάνες θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερο από το 2% και άρα προκύπτει το ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν έτσι να τηρηθούν αυτά τα οποία δηλαδή είχε δεσμευτεί να κάνει πριν από λίγα χρόνια ο κύριος Μπαρόζο αυτό το οποίο είναι ενισχυτικό είναι πως η ίδια η Κομισιόν παρατηρεί πως ε, τα ποσά αυτά ε, δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Ειδικά όσον αφορά την πολιτική συνοχής γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες ε, επιφυλάξεις οι οποίες εκφράζονται και είναι κάπως δύσκολο να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Να γίνω πιο συγκεκριμένο στο τομέα της γεωργικής ανάπτυξης. Μας λέει το ελεγκτικό συνέδριο πως έχουμε ποστό του 7,7% το υψηλότερο στην κοινωτική πολιτική και λέει πως θα είναι αδύνατον να έχουμε σημαντική επίδραση τώρα στο ποσοστό σφάλματος φέτος ή του χρόνου. Οπότε έτσι η Κομισιόν θεωρώ αναγνωρίζει πως τα μέτρα αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα οδηγήσουν σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα σε ε, κάποιο σε κάποιον άμεσο όριζοντα. Οπότε θα ήθελα εγώ να σας ζητήσω να αναβάλουμε τη διαδικασία απαλλαγή ή δεν ξέρω τι θα μπορούσε να μας προτείνει η Κομισιόν και να μας συστήσει γιατί δεν ξέρω αν μπορούσε να προτείνει κάτι άλλο κατόπιν ένα άλλο ζήτημα που αφορά τη Γενική Διεθνή Συριακή Α, εκεί πέρα μας λέει η Κομισιόν πως θα πρέπει να υπάρξει μια επικαιροποίηση της διαδικασίας. Ε, θα θέλαμε να μάθουμε αν έλαβε μια απόφαση το σώμα των επιτρόπων σχετικά και αν ναι, ποιες, ποια είναι τα κύρια σημεία αυτής της απόφασης. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ κύριε Πίπερ. Κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ που ήρθατε κυρία Γενική Γραμματέα. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα 1 του ερωτηματολογίου, δηλαδή το γιατί οι απαντήσεις των επιτρόπων περιορίστηκαν σε 25 σελίδες. Είναι ζήτημα λογοδοσίας. Και το επόμενο ερώτημα είναι το γιατί δεν ασχολήθηκε το σώμα των επιτρόπων με αυτό. Στην απάντηση αναφέρεται πως ε, το γκρι η διοργανική ομάδα δηλαδή όπως λέγεται δεν ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα. Ε, οπότε έχουμε πολιτικά ζητήματα και εδώ πέρα κάποιοι ε, τεχνικοί μας λένε τι πρέπει να γίνει. Ε, δεν είναι δυνατόν. Και δεν ε, ανέβηκε και στην εκτίμησή μου η Επιτροπή που συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Ασχολήθηκε λοιπόν το Σώμα των Επιτρόπων. Εάν δει επίσης κανείς τα νούμερα πρέπει να πούμε πως πάρα πολλά ε, κοινοβουλευτικά ερωτήματα ενδιαφέρουν τους ψηφοφόρους μας. Να καταλαβαίνω πως κάποια πράγματα είναι κουραστικά και δεν είναι δυνατόν να απασχολούν την Επιτροπή, αλλά κάποια άλλα ζητήματα δεν είναι σημαντικά και δεν έχουν απαντηθεί καθόλου ικανοποιητικά. Και το ερώτημα τι αξίζει αυτή η διαδικασία και τι ε, νόημα έχει τελικά η διαδικασία της λογοδοσίας δεδομένης δεδομένων αυτών των απαντήσεων. Επίσης, ένα ζήτημα που είναι δική σας ευθύνη, εξέταση Βουλγαρίας και Ρουμανίας όσον αφορά τη μεταρρύθμιση δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εάν δούμε ε, την διεθνή διαφάνεια η οποία εκτιμά πως η Βουλγαρία από τη θέση 64 έπεσε στη θέση 77 υπό την επιτήρηση της Κομισιόν και η δε Ρουμανία δεν μετακινήθηκε από τη θέση 69 της παγκόσμιας διάφορας. Δεν θεωρώ πως είστε και τόσο επιτυχημένοι. Εσείς πώς αξιολογείτε τη διαδικασία και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να γίνουν πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε και ικανοποιημένοι με την κατάσταση στις χώρες αυτές. μια πίσω πως δεν βελτιώνονται τα πράγματα. Θα ήθελα μια απάντηση λοιπόν. Νομίζω αξίζουμε μια τέτοια απάντηση. Έχουμε τη 13η έκθεση πλέον. Γι' αυτό παρακαλώ μια απάντηση. Επίσης καλό θα ήταν να μάθουμε πότε θα λάβουμε απαντήσει στα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε θέσει. Και το τέταρτο αφορά συμβάσεις χωρίς διαγωνισμό. Έχουμε πολλές διαπραγματευτικές διαδικασίες χωρίς... Έχουμε πολλές ε, συμβάσεις, με χωρίς ε, κάποια... κάποιο διαγωνισμό. Αυτό θα ήθελα να το κάνουν και κάποιοι δήμοι και κάποια μέλη αν μπορούσαν, έτσι. Βλέπουμε εδώ πέρα 40 εκατομμύρια μελέτη ε, του συστημάτων δικαιοσύνης 200.000 ευρώ. Γιατί δεν κάνετε ένα διαγωνισμό. Δεν θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Ευχαριστώ Γιάννη Μούλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κομισιόν στην εισαγωγή της έδωσε βάρος στην απλούστευση των διαδικασιών. Κάτι το οποίο συνδιαφέρει την Επιτροπή μας, νομίζω όλοι είναι υπέρ και γι' αυτό τον λόγο πριν από κάποια χρόνια ε, λάβαμε την πρωτοβουλία πως ε, πρέπει να γίνει κάτι. Αυτό το οποίο λέμε δηλαδή είναι ομάδα Στόιμπερ, ε, η θητεία της οποίας όμως θα τελειώσει στο τέλος του έτους. Θα ήθελα να γνωρίζω ποιε είναι οι προθέσεις, ποια είναι η εμπειρία της Κομισιόν με την ομάδα στο μέχρι και αν έχει κάποια πρόθεση η Κομισιόν να προτείνει να συνεχιστεί η δουλειά της. Ε, και το άλλο ερώτημα που ανακύπτει συχνά. Στο τέλος του θα έχουμε νέα κομισιόν. Θα διαλυθούν τα γραφεία των επιτρόπων και οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε ως ελεξιωτιστές σε διάφορες θέσεις. Πώς διασφαλίζετε την δικαιοσύνη στις προαγωγές και να μην ε, ευνοούνται μόνο αυτοί που δούλευαν στα γραφεία των επιτρόπων, αντί για τους κανονικούς υπαλλήλους της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Μπάρτ. Μπάρτ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ Σας καλωσορίζουμε κυρία Ντέι. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε θέσει και στη ερωτηματολόγια όσον αφορά τις ε, περιστρεφόμενες πόρτες εκεί πέρα μεταξύ διαφόρων αξιωμάτων. Στην, ε, επιτροπή, στην προηγούμενη επιτροπή Μπαρόζο είδαν πως ε, έφυγαν κάποιοι 13 νομίζω επιτροποί, 6 από αυτούς ε, πήγαν στον ιδιωτικό τομέα ε, και στα λόμπι. Και θεωρώ κυρία Ντέι πως η Κομισιόν παρακολουθεί με το τι κάνετε για να ρυθμίσετε καλύτερα το ζήτημα γιατί η Κομισιόν λέει συνέχεια πως η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κρίνει το εάν και πως μπορούν να συνεχίσουν τι δραστηριότητε τους κάποιοι επιτροπή. Μήπως θα έπρεπε τώρα να ξεκαθαρίσουμε το τι γίνεται συγκεκριμένα με το θέμα αυτό, το τι επιτρέπεται, το τι απαγορεύεται και το τι απαγορεύεται αυστηρά ένα άλλο θέμα στο ερωτηματολόγιο για τους επιτρόπους. Ε, Είπαμε πως υπάρχει μία περίοδος ηρεμίας η οποία προβλέπεται. Βλέπω εδώ πέρα στις ε, ερώτηση 41 πως ανέβηκε από τους 12 μήνες στους 18 αλλά βλέπω πως έχουν και ένα επίδομα ε, για τρία χρόνια. Μήπως θα έπρεπε και το επίδομα να είναι 18 μήνες ε, έτσι, γιατί αν υπάρχει μία περίοδος ε, ηρεμίας στην οποία δεν επιτρέπεται να αναλάβουν άλλα καθήκοντα η οποία δεν αρκεί 18 μήνες νομίζω ότι αρκεί και το επίδομα που δίνεται στους αποχωρούντες επιτρόπους να διαρκεί τόσο. Τρίτη ερώτηση. Τέσσερις έχω σύνολο. Η Επιτροπή Ηθικής ε, που πρέπει να είναι επαγγελματική και ανεξάρτητη. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποια προβλήματα με τον Μισελ Πετή, ο οποίος ε, είχε δραστηριοποιηθεί και στην Επιτροπή Ελέγχου του Υπερπολογισμού και εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα για την ανεξαρτησία του, γιατί βεβαίως εργάζεται και σε ένα δικηγορικό γραφείο. Τα γνωρίζετε αυτά. Τέλος πάντων συνέβη ό,τι συνέβη, αλλά τώρα η στην ερώτηση 36 απαντάει ε, πάρα πολύ χαλαρά. Δηλαδή η διαμεσολαβήτρια είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και εσείς πολύ απλά λέτε δεν συμφωνούμε με αυτά τα οποία είπε η διαμεσολαβήτρια. Γιατί. Ε, έκανε κάποιες πολύ έντονες ε, δηλώσεις και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ακούσουμε την άποψή σας. Και ένα άλλο ερώτημα το οποίο φαντάζομαι δεν μπορείτε να το απαντήσετε τώρα, αλλά θα ήθελα να το απαντήσετε γραπτός. Στο παράρτημα που αναφέρεται στις συμβάσεις εξωτερικών συμβούλων. Αναφέρεται μια εταιρεία Bows Company. Έλαβε 198.000 ευρώ. BOZ. Boson Company. 198.000 λοιπόν ευρώ. Εγώ θα ήθελα να μάθω τι ε, συμβουλές έδωσε αυτή η εταιρεία. Ένας από τους εργαζόμενους της εταιρείας ο κύριος, ήταν ο κύριος Σνόντεν. Έτσι, εργαζόταν για την Bose Company και έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εταιρεία αυτή 108.000 Ξέρω Φαντάζομαι πως δεν μπορείτε να απαντήσετε τώρα αμέσω. Αναμένω όμως μια ε, γραπτή απάντηση. Ευχαριστώ. Αυτές ε, είναι οι ερωτήσεις μου κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεγιόν είναι τελευταίος στον κατάλογο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Γενική Γραμματέα, την κυρία Ντέι. Νομίζω όλοι θέλουμε να έχουμε ένα σωστό διάλογο εδώ πέρα στις περιπτώσεις αυτές, θετικό αυτό όσον αφορά το έγγραφο αυτό Να αναφερθώ πρώτα απ' όλα 46 για τους πληροφοριοδότες. Ζητάμε μια αξιολόγηση από την Κομισιόν για το πώς λειτουργεί τώρα το σύστημα και η απάντηση είναι πως είχαμε κάποια κατάρτιση, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να μάθουμε είναι οι εργαζόμενοι της Κομισιόν που αφορούν τα ζητήματα ηθικής έχουν κάνει τίποτα ή όχι. Έχουν λάβει ανώνυμες καταγγελίες. Για αυτό το οποίο είπε ο Μπαρτστάς συμφωνώ μαζί του για τα αξιώματα και την αναλλαγή αξιωμάτων. Μετά υπάρχει μια δύσκολη συζήτηση για την αξιολόγηση αντικτύπου, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα ερωτήματα που ε, υπάρχουν εδώ πέρα. Αλλά ε, υπάρχουν πάρα πολλά μπορεί στην απάντηση της Κομισιόν. Μπορεί να υπάρξει συνέχεια, μπορεί να οφείλεται η αντίδραση του Όλαφ σε αυτό, μπορεί να οφείλεται στο άλλο. Είναι μάλλον απίθανο να γίνει δεκτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από όλα τα κράτη-μέλη, οπότε θα έχουμε και τον Όλαφ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα λειτουργούν σε κάποια μόνο κράτη-μέλη. Με βάση αυτά, εγώ, εάν ήμουν στη θέση της Κομισιόν, θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να βελτιώσω τον Όλαφ ε, και την ποιότητα των ερευνών του έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα επικοινωνίας και να υπάρχει κάποια συνέχεια από πλευρά καθών μελών. Συμφωνείτε λοιπόν πως πρέπει να έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό από όλα αυτά τα μπορεί και τα ίσως από πλευρά Κομισιόν. Μετά σελίδα 26. Απογοητεύομαι λίγο από την απάντηση της Κομισιόν όταν ε, μιλάμε για τη μελέτη του επίπεδου πληρωμών. Η Επιτροπή Έλεγχου του Προπολογισμού το 2012 ζήτησε μια σχετική μελέτη και μας είπατε πως η Κομισιόν δεν το θεωρεί αναγκαίο γιατί τώρα έχουμε νέους κανόνες για το προσωπικό. Αλλά μπορώ να σας πω πως στο επίπεδο των πολιτών ε, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς εξηγείται τη διαφορά ε, εθνικών μισθών και κομισιών. Και εάν θέλετε, νομίζω, περισσότερη στήριξη από τους πολίτες για την εξτάμενη κατάσταση, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια τέτοια μελέτη. Και το επιχείρημα πως δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να δώσουν τις πληροφορίες, ε, νομίζω μπορεί να λυθεί. Μπορεί να σας βοηθήσει το Κοινοβούλιο να λάβετε τις πληροφορίες. Μετά, σελίδα 30. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες Είχαμε χθε μια ακρόαση. Πρέπει να λυθούν κάποια οριζόντια ζητήματα, π.χ. για την Επιτροπή μας. Έχουμε κάποιες προφορίες όχι τόσο καλές. Έχουμε κάποιες γενικέ κατευθυντήριες γραμμές, αλλά εγώ θα ήθελα να δούμε για την, με την εφαρμογή του το τι γίνεται. Δηλαδή, θα ήθελα η Κομισιόν να διευνήσει πού πάνε καλά τα πράγματα, πού πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή και ανησυχώ από την παρατήρηση που υπάρχει εδώ πέρα. Πώς οι υπηρεσίες αυτές είναι νομικά ανεξάρτητες και είναι οι μόνες υπεύθυνε ε, για το πώς ε, θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό στην πράξη. Όχι, η Κομισιόν έχει την εποπτεία των ε, οργανισμών αυτών. Αλλιώς υπάρχει κάποιο κενό, έτσι. Τέλος, για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, συμφωνώ. Ως πρόεδρος ε, μιας ομάδας ε, ευρωβουλευτών για το ότι έχουμε νομίζω μια καλή επαφή αλλά δεν αντιλαμβάνουμε την άρνηση της Κομισιόν να ζητήσει από τις γενικές διευθύνσεις να αντιδράσουν γιατί μας παρέπεμψε ο Γενικός Γραμματέας στις γενικές διευθύνσεις οπότε νομίζω πως λογικό είναι να ρωτήσουμε από τις γενικές διευθύνσεις να δώσουμε μια απάντηση γιατί εκεί μας παραπέμπει η Γενική Γραμματέας Μάλιστα ε, Έχουμε πολλές ερωτήσεις Κύριε Αντέη, παρακαλώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις με τη σειρά που ακούστηκαν. Όσον αφορά την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία διακυβεύονται και για ποιο λόγο έχουμε ξεπεράσει το 2% όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σφάλμα δεν σημαίνει απαραίτητα απάτη, το σφάλμα ως έννοια καλύπτει πολλά διαφορετικά πράγματα. Επομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μειωθεί προφανώ ο αριθμός των σφαλμάτων και γι' αυτό ακριβώ το λόγο επιμείναμε πάρα πολύ στο ζήτημα τη απλούστευση. Πάρα πολλά σφάλματα προκύπτουν από αρχέ τη αυτοδιοίκηση που δεν είναι σε θέση πολλέ φορέ να καταλάβουν τι ακριβώ πρέπει να κάνουν και προσπαθούν ουσιαστικά να ανταποκριθούν σε κάποιους κανόνες πολλέ φορέ είναι και πολύ πολύπλοκοι. Ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά και το ξέρει και η δική σας Επιτροπή ότι κατά τη διάρκεια του κύκλου του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου ξέρετε ότι έχουμε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό σφάλματος στην αρχή της περίοδου ακριβώς επειδή τα έργα δεν έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται και με την ολοκλήρωσή τους βέβαια το ποσοστό αυτό σφάλματος αυξάνεται και έτσι καταλήγουμε και στα ποσοστά που τα οποία έχουμε για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Αυτό το οποίο εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να καταφέρουμε να ενισχύσουμε ενισχύσουμε τους ελέγχους όπου ήταν δυνατό. Είμαστε εμεί υπεύθυνοι για την άμεση διαχείριση ένα μικρού ποσοστού του κοινοτικού προπολογισμού, το 80% του κοινοτικού προπολογισμού αποτελεί αντικείμενο επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν στο εφιστάμενο πλέον δημοσιονομικό πλαίσιο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πλέον μία προσέγγιση η οποία είναι πιο ολοκληρωμένη και πιο σφαιρική σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο, όσον αφορά δηλαδή τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ απαιτητικοί και ασκήσαμε πίεση στα κράτη-μέλη χρησιμοποιώντας εργαλεία, μέσα όπως η διακοπή, αναστολή των κοινοτικών δαπανών. Σας πεθυμίζω πάντως ότι για ένα 80% του κοινοτικού προπολογισμού έχουμε κοινή διαχείριση με τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του χρόνου που απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθούμε σε κάποια ερωτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αύξηση των δαπανών σε πάρα πολλού τομεί, το γεγονό ότι πρέπει να κινητοποιηθούν πάρα πολλοί πόροι. Καταλαβαίνω επίση ότι οι απαντήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μεταφραστούν σε όλε τι επίσημε γλώσσε Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί στο σύστημα διαλόγου που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε πάνω από 13.000 ερωτήσεις που μας έρχονται κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις αυτές και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στην κάθε μία ερώτηση όσο πιο σφαιρικά γίνεται. Αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές αναγκαζόμαστε να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις μας θέτατε ερωτήσεις και εμείς επαναλαμβάναμε τις απαντήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα λίγο πιο αποτελεσματικό, λίγο πιο ευσύνοπτο. Να μπορούμε δηλαδή να απαντάμε άμεσα σε κάποιες ερωτήσεις, ολιγόλογα, χωρίς να γράφουμε ολόκληρη έκθεση κάθε φορά. Επίσης νομίζω ότι πάρα πολλές ερωτήσεις θα μπορούσαν να απαντηθούν με την παροχή περαιτέρων πληροφοριών, με την παροχή κάποιων παραρτημάτων. Μπορείτε άμεσα δηλαδή εσείς σε κάποια επιπλέον έγγραφα να βρείτε τις απαντήσεις τις οποίες θέλετε. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα ερωτήσεων και απαντήσεων και με άλλε επιτροπέ και τμήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθούμε να δούμε πώ μπορούμε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθούμε στον αυξανόμενο αριθμό κοινοβουλευτικών ερωτήσεων που μα φτάνουν σε αιτήσια βάση. Το Σώμα των Επιτρόπων προφανώ λαμβάνει υπόψη του τα συμπεράσματα της ομάδας GRIP είναι η ομάδα αυτή η οποία ασχολείται με τα διοργανικά ζητήματα, ουσιαστικά με τη συνεργασία που έχουμε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και όπως σας λέω και στην απάντησή μου, το σώμα των επιτρόπων έχει συμφωνήσει με τη διαδικασία αυτή όταν άρχισαν να ισχύουν οι νέοι αυτοί κανόνε. Για το CPM πρέπει να σα πω, και το λέω και στην κυρία Γκρέσλερ και στου υπόλοιπου, ότι αύριο το σώμα των επιτρόπων θα εγκρίνει νέε εκθέσει όσον αφορά το μηχανισμό CVM για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Επομένω θα έχετε τις νέες αυτές εξελίξεις και τη νέα αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δύο αυτές χώρες ήδη αύριο. Ξέρετε ότι είναι μακροσκελή η διαδικασία αυτή, δεν αλλάζουμε απλώς το νομικό πλαίσιο, στα πλαίσια του οποίου το κράτος δικαίου εφαρμόζεται σε αυτά τα κράτη-μέλη, αλλά τροποποιούμε επίσης και την ίδια την οτροπία των ανθρώπων, των υπευθύνων για τα διάφορα προγράμματα. Οι δύο αυτές χώρες προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Δεν έχουμε λοιπόν τον ίδιο αριθμό εκθέσεων όπως για τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως στις 6-7 εκθέσεις που έχουμε υποβάλει προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στις χώρες αυτές και για το πώς μπορούν οι χώρες αυτές να έχουν ε, ένα καλύτερο σύστημα παρακολούθησης του δικαστικού τομέα και πώς μπορούν επίσης να παρακολουθούν καλύτερα τις αλλαγές που γίνονται σε κάποιες νομοθεσίες. Θα αναφερθώ εκτενέστερα στις, στα ζητήματα αυτά στις εκθέσεις τις οποίες θα λάβετε αύριο. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των συμβάσεων χωρίς πρώτερο διαγωνισμό, νομίζω ότι σας έχουμε δώσει ιδιαίτερα λεπτομερείς απαντήσεις. Σας εξηγούμε πώς συνέβη το κάθε τι. Σε ορισμένες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί κάποιες διαδικασίες διαπραγμάτευσης, εκεί δηλαδή όπου έχουμε χαμηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης εκεί όπου ενδεχομένως να έχουμε ακόμα και μονοπόλιο όσον αφορά τους προμηθευτές, επειδή ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο ζήτημα προστασίας δικαιωμάτων πνευματικών ή δικαιωμάτων του δημιουργού ή σε τομείς όπου απαιτούνται πολύ εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις. Ή μερικές φορές έχουμε συμβάσεις χωρίς διαγωνισμούς για περιπτώσεις όπου υπάρχει αποκλειστικότητα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση κάποιων πνευματικών δικαιωμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε δημόσιο διαγωνισμό για λόγους ε, αποτελεσματικότητας για λόγους εξοικονόμησης. Θα ήταν παράλογο άλλωστε να κάναμε κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω ότι από καιρού εις καιρών προκύπτουν κάποιες έκτακτες περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι η απάντησή μου πρέπει να σας καλύπτει. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Μούλτερ για την απλούστευση, απλοποίηση. Ναι, όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ζήτημα της βελτίωσης της νομοθεσίας μας και αυτό καλύπτει μια μεγάλη γάμα δραστηριοτήτων το σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας για παράδειγμα και πώς αξιολογείται αυτό σε διάφορες προτάσεις που κάνουμε, αλλά καλύπτουμε επίσης και το σύνολο της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας. Θα γνωρίσετε το πρόγραμμα REFIT, καθώς επίσης και τη σχετική ανακοίνωση πέρυσι το φθινόπωρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου ε, αναφερθήκαμε σε πολλά πολυετή προγράμματα που θα μας επιτρέψουν να ελέγξουμε κάθε κοινοτική νομοθεσία, να δούμε αν πραγματικά ανταποκρίνεται πλέον στις περιστάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις θα γίνουν βελτιώσει προσαρμογές, σε άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως να καταργήσουμε και να αποσύρουμε κοινοτική νομοθεσία ή να οδηγηθούμε ακόμα και στην κατάργηση κάποιων νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα Stoiber είναι μια συμβουλευτική ομάδα στην οποία συμμετέχουν διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπρόσωποι του βιομηχανικού τομέα, εκπρόσωποι εθνικών φορέων. Όπως είπε και ο κύριος Μούλτερ, η εντολή της ομάδας αυτής ολοκληρώνεται στα τέλη του 2014 δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να κάνω προβλέψεις για το πώς θα αντιδράσει η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά φαντάζομαι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα επιθυμήσει να συνεχιστεί το έργο αυτό που κάνει η ομάδα Στόιμπερ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να επεμβαίνει μόνο στο σωστό επίπεδο και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Είναι σημαντικό να επεμβαίνουμε με τον πιο ήπιο τρόπο και θα πρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορούμε πραγματικά να ελέγχουμε την νομοθεσία την οποία εφαρμόζουμε. Πράγματα τα οποία ισχύουν για τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια ενδεχομένω να μην ανταποκρίνονται πλέον στι πραγματικέ ανάγκε Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά το γενικότερο πρόγραμμα βελτίωση τη νομοθεσία έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική αξιολόγηση πολλές φορές και εκ των προτέρων για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί η κοινοτική νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή προχωράμε σε μια αξιολόγηση εκ των υστέρων, εξ και επιθυμούμε πολλά κράτη-μέλη να συνταχθούν με το δικό μας ε, το έργο, όσον αφορά δηλαδή την αξιολόγηση της νομοθεσίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αυτό έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αξιολογήσεις αντικτύπου, όσον αφορά πάντα την κοινοτική νομοθεσία και εμείς προφανώς αυτό το στηρίζουμε. Πάντως, σας έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν νομοθετεί το Συμβούλιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να αρχίσει να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο αξιολογήσεις αντικτύπου. Αυτό αναμένουμε λοιπόν από το Συμβούλιο, αυτό περιμένουμε από το Συμβούλιο, αλλά περιορίζομαι, αν θέλετε, μόνο σε αυτό τον ευσεβή πόθο. Και ελπίζω ότι και η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει αυτή την προσέγγιση. Θα πρέπει όλοι ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε αν η κοινοτική νομοθεσία μας και αν οι επιμέρους πολιτικές όντως αποδίδουν αποτελέσματα και αν όχι θα πρέπει να διορθώνται και να προσαρμόζονται. Όσον αφορά τώρα το τελικό αυτό στάδιο της θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στα γραφεία των επιτρόπων θα αρχίσουν να απασχολούνται μετά το τέλος της θητείας αυτής σε άλλες διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προφανώς εδώ πέρα ακολουθείται η ε, κλασική παραδοσιακή διαδικασία. Κοιτάξτε, ο όρος revolving doors, περιστρεφόμενες πόρτες, δεν μ' αρέσει πολύ. Αναφέρομαι σε αυτή την μεταπίδηση στην οποία αναφερθήκατε στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε ότι υπάρχει για τους επιτρόπους ένας κώδικας συμπεριφοράς και δεντολογία. Επικαιροποιήθηκε μάλιστα πρόσφατα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματικά εφαρμόζει τέτοιους κανόνες δεντολογία. Είμαστε λοιπόν πολύ αυστηροί και θα θέλαμε να δούμε και τα άλλα θεσμικά όργανα κάνουν κάτι ανάλογο. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε καταφέρει να συσπίσουμε αρκετά, νομίζω. Ε, Πάντω τονίζομαστε οι μόνοι που ακολουθούμε του κανόνε αυτού. Όσον αφορά αυτή την περίοδο ηρεμία στην οποία αναφέρθηκε ο κύριο Στά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνη τη αποφάσισε να επιμηκυνθεί στου 18 μήνε από 12. Τώρα, όσον αφορά τα σχετικά επιδόματα, υπάρχουν συγκεκριμένα νομικά κείμενα τα επιδόματα αυτά δίνονται για τρία χρόνια, αφού τα αποχωρήσει από την Επιτροπή ένας Επίτροπος. Ορισμένοι δεν απασχολούνται σε κάποια άλλη εργασία στη συνέχεια επαμοιβή, άλλοι πάλι το κάνουν. Πάντως σε κάθε περίπτωση σταθμίζουμε έτσι την κατάσταση ώστε να επιτρέπουμε στους επιτρόπους να βρουν μια άλλη απασχόληση εφόσον το επιθυμούν μετά το τέλος θητείας τους. Πολλοί άλλωστε επίτροποι είναι αρκετά νέοι, επομένως επιθυμούν προφανώς να απασχοληθούν σε κάποια άλλη θέση στο μέλλον. Και υπάρχουν πάντως πολύ συγκεκριμένοι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους εφόσον στην τριετή αυτή περίοδο βρουν μια άλλη εργασία, οι αποδοχές τους ή μάλλον το επίδομα το οποίο παίρνουν κατά την περίοδο ηρεμίας προσαρμόζεται ή μειώνεται με βάση το μισθό που αρχίζουν να παίρνουν στη νέα θέση απασχόλησής τους. Και όσον αφορά και την ad hoc Επιτροπή Διοντολογίας, τα μέλη της Επιτροπής αυτής είναι ανεξάρτητα, κανείς δεν τους υποδεικνύει πώς θα πρέπει να αποφασίζουν ή τι αξιολογήσεις θα πρέπει να κάνουν. και θεωρούμε ότι αυτή η ad hoc Επιτροπή διοντολογία επιτελεί ένα πολύ σωστό και επαγγελματικό έργο, χωρίς να πειράζεται δηλαδή από υφιστάμενους ή πρώην επιτρόπους. υφιστάμενου η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μία απόφαση για το αν θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένα πρότυπα ξεχωριστά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το έργο των Επιτρόπων. Όσον αφορά την επόμενη ερώτηση του κ. Στάς, δεν μπορώ αυτή τη απαντήσεις, θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες αργότερα. Όσον αφορά τώρα πάλι την Επιτροπή αυτή ιδεντολογία. ουσιαστικά, μάλλον όσον αφορά τους πληροφοριδότες, με συγχωρείτε, ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί επιθυμούν να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου κάθε φορά που εντοπίζουν κάποια προβλήματα. Ξέρετε ότι έχουμε και μία εβδομάδα αφιερωμένη σε ζητήματα διοντολογία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθούμε να προωθούμε μέσω τη εβδομάδα αυτή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πέρα από τι άλλε αρμοδιότητε που έχουν άνθρωποι αυτοί με τη συμμετοχή του στην ομάδα, την Επιτροπή Διοντολογία, ασχολούνται και με τα ζητήματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενθυμίζουμε σε όλου του εργαζομένου Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε και ότι αυτοί θα πρέπει να τηρούνται. Και αυτό το κάνουμε με την υποβολή συχνών ερωτήσεων, με το να προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις σε κάποιες υποθετικές ερωτήσεις, σε κάποια υποθετικά σενάρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τι επαιτούμε από αυτούς. Όσον αφορά τώρα την Όλαφα και το ζήτημα του EPPO, νομίζω ότι ήδη έχουμε απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας νέος κανονισμός για το καταστατικό της Όλαφα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε και μία σχετική ανακοίνωση για το πώς μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο η λειτουργία της Όλαφ από διάφορες πτυχές. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο έχουμε θέσει επιτάπητος για περαιτέρω συζήτηση και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια μαθητική πρόταση προκειμένου να διασφαλίσει τις ε, ίδιες ε, εγγύησεις με αυτές που ισχύουν για την υπόθεση PPO. Να ισχύουν δηλαδή οι ίδιες απαιτήσει και για την Όλαφά. Όσον αφορά τώρα το επίπεδο αποζημιώσεων, νομίζω ότι είναι κάπως σύντομη η απάντηση. Πάντως στην όλη συζήτηση και στις διαπραγματεύσεις που είχαμε για την μέθοδο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να καταρτιστούν οι μελλοντικές αποδοχές για τους εργαζομένους, εμείς δώσαμε πάρα πολλές πληροφορίες για τους διεθνείς οργανισμούς, για το τι γνωρίζουμε για τα κράτη-μέλη στα οποία αποσπώνται μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν γίνει λοιπόν ενδελεχείς υπολογισμοί. Συμφωνώ μαζί σας ότι αν οι Ευρωπαίοι θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλέ πληροφορίες, είναι δημόσιες και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να εξηγήσουμε περισσότερο πώ διαμορφώνονται οι μισθοί σε κάθε χώρα. Νομίζω πάντω ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη αποφασίσει για το πώ θα υπολογίζονται οι μισθοί στο μέλλον και ελπίζω ότι η μεγαλύτερη αυτή προσοχή που θα δοθεί στο επίπεδο των μισθών στο μέλλον θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει, να έχουμε πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Όσον αφορά τώρα τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την λειτουργία των οργανισμών αυτών. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά μαζί τους, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους οργανισμούς αυτούς, πολλοί εκ των οποίων είναι πολύ μικροί. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε μέσω πυρογνωμοσύνης ε, κάποιους οργανισμούς ε, σε ζητήματα διαχείρισης και λειτουργίας, αλλά είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι, τα διοικητικά του συμβούλια δηλαδή, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Εμείς προσπαθήσαμε να καταρτήσουμε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για τη σύγκρουση συμφερόντων και μετά από κάποιο καιρό, αφού τους αφήσουμε δηλαδή λίγο χρόνο, θα κάνουμε και μία έρευνα για να δούμε πώς εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις αυτές γραμμές από τους ε, εξωτερικούς αυτούς αποκεντρωμένους οργανισμούς. Επαναλαμβάνω πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι άμεσα υπεύθυνη για τον τρόπο λειτουργία τους. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι κάλυψα όλες τις ερωτήσεις, διαφορετικά θα ξαναπάρω το λόγο. Ε, ε, ευχαριστώ. Δύο συνάδελφοι έχουν ερωτήσεις, Κρέσλε και Πίπερ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ θα ήθελα να έχω μια ημερομηνία για το πότε υποβλήθηκε η απόφαση του Γκρι στους επιδρόχους. για να περιοριστούν οι απαντήσεις σε 25 σελίδες. Μετά, κυρία Αματέα, λέτε πως μπορεί να απαντήσει κανείς σε 25 γραμμές. Ναι, αλλά όχι όλα, όχι τα πάντα, δεν λύνονται όλα σε 25 γραμμές. Μπορώ να σου πω πολλά παραδείγματα. Ε, δεν αφορούν ε, κάποιο, κάποια συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, αλλά θεωρώ πως ε, χάνει μια ευκαιρία εδώ πέρα η Κομισιόν για να απαντήσει αξιοπρεπώς. Λέτε πως μπορεί να απαντήσει κανείς τα παραρτήματα. Ναι, αλλά τα παραρτήματα δεν μπαίνουν στο ίντερνετ, δεν είναι δημόσια. Εσκεμένα. και δεν είναι σίγουρο πως θα λάβει κανείς απάντηση και στα παραρτήματα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω πως επιμένω πως είναι βήμα προς τα πίσω και δεν θεωρώ πως είναι σωστό να περιοριστεί η λογοδοσία. Μετά Βουλγαρία, Ρουμανία. Εντάξει, θετική η αυριανή έκθεση, αλλά Μια έκθεση δεν μου λέει τίποτα εμένα. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε για να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία λέει η έκθεση. Η ε, αμνηστία στους πολιτικούς ε, της Ρουμανίας ε, οι οποίοι παρόλη τη διαφθορά θα είναι ελεύθεροι δεν μπορούμε τότε να συνεχίσουμε να τους δίνουμε λεφτά. Έχουμε πολλές εκθέσεις ήδη. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κρέσλε. Κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ. Απαντήσατε εν μέρη στα δικά μου τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Το ερώτημα ήταν τι γίνεται με αυτή την αξιολόγηση του κινδύνου, αν ε, σημαίνει κάτι αυτό για μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Και μετά δεν απαντήσετε και άλλη μια ερώτηση που αφορά τα διαδικαστικά λάθη στην και το βαθμό σοβαρότητάς τους ε, στην ε, πολιτική συνοχή. Υπήρξε νομίζω μια απόφαση της Κομισιόν για επανακαθορισμό ακριβώς του σοβαρού βαθμού λάθους και τελευταίο Είπατε πως στην Κομισιόν έχουμε αυστηρούς κανόνες, έχουμε έναν κώδικα συμπεριφοράς τον οποίο τηρούμε και μας το γράψατε όλα σε αυτό. Επίσης έχετε και εσωτερική υποχρέωση στην Κομισιόν για να υπάρχει εναλλαγή των στελεχών ε, των διευθυντικών κάθε πέντε χρόνια και αυτό νομίζω ισχύει και για τα ανώτατα αξιώματα. Θα ήθελα να μάθω τι γίνεται και με εσάς προσωπικά λοιπόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ντέι, μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον, όσον αφορά το τι απάντηση πρέπει να δίνετε σε μια κοινωνική ερώτηση. Πόσο μακρά πρέπει να αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη το τι συζητάτε, οπότε το, τότε που είπατε το Σεπτέμβριο του 2011, τότε εμείς ε, λάβαμε γνώση και συμφωνήσαμε. Τώρα αφορά τις απαντήσεις. Ακόμα δεν μας έχει υποβληθεί μια ερώτηση που δεν μπορεί να τύχει απαντήσει 25 στίχους. Δεν είναι tweet, που να σε πετάει έξω από το σύστημα εάν υπερβείς τους χαρακτήρες που επιτρέπονται. Τέλος πάντων έχουμε λιγότερες εξαιρέσεις και ό,τι χρειάζεται τα συζητούμε και πάντοτε βρίσκουμε έναν τρόπο να είμαστε συγκεκριμένοι και ευσύνοπτοι. Επομένως, είναι δυνατόν να υπερβούμε το σχετικό όριο, αλλά δεν χρειάζεται. τόσο πάντων δεν μπορώ να το αποκλείσουν τι θα συμβεί κάτι. Τόσο αφορά και Βουλγαρία και την Ρουμανία. Ο μηχανισμό αυτό συνεργασία και επαλήθευση. Αυτό θα το κάνουμε. Βοηθήσουμε τι χώρε όσον αφορά το δύσκολο έργο του. Και άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον ε, μηχανισμό. Θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και εξωτερική βοήθεια άρχισε να στις στατιστικές του Ευρωβαρομέτρου ε, τι γίνεται για αυτού που διαμαρτυρούνται τόσο καιρό στη χώρα, στη Βουλγαρία σημαίνει ότι υπάρχει διακαεί πόθο από πλευρά του κόσμου τη χώρα αυτές Ούτω ώστε να υπάρξει εξηγήση της δικαιοσύνη, ε, και τη κρατική μηχανής γενικότερα να πλησιάσουν περισσότερο τα κοινοτικά πρότυπα. Νομίζω ότι κάνουμε ένα έργο το οποίο είναι απαραίτητο και δύσκολο. Βοηθούμε τις κυβερνήσεις των χρόνων αυτών και σιγά σιγά οι προσπαθειές μας αποδίδουν. Όπως σας είπα, έχει αλλάξει όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά Βλέπετε αλλαγέ και στους δικαστές και σε όλου του εμπλεκομένου. Αλλαγή Θέλουν πολύ να πλησιάζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πάντως αυτά δεν αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Και το θέμα δεν είναι κανείς να κάνει νομοθετική μεταρρύθμιση, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία σε όλη την κλίμακα των εμπλεκομένων και του κόσμου. Κύριε Πίπερ, δεν ξέρω αν κατάλαβα 100% την άλλη σας ερώτηση. Να σας, σας απαντήσω πάνω σε αυτό που κατάλαβα. Νομίζω ότι ρωτήσατε για το κατά πόσο θα πρέπει να έχουν επιφυλάξει οι γενικοί διευθυντές όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος. Ναι, ο καθένα, πάντω αναλαμβάνει τι ευθύνε του ε, σε σχέση με το τι επιφυλάξει θα διατυπώσει. Θα πρέπει κάθε γενική διεύθυνση να σταθμίσει πώς διακυμαίνονται ή πώς αυξάνεται το ποσοστό σφάλματος. Τα συζητήσαμε χρόνια και με το ελληνικό συνέδριο. Δεν συμφωνήσαμε σε όλα. Από την εμπειρία πάντως ξέρουμε ότι 2% είναι πολύ χαμηλό, ε, Λαμβάνοντα υπόψη και το κόστος των ελέγχων είναι καλό σαν στόχος. Δεν γίνεται σε όλους τους τομείς να έχουμε 2% ή τέλος πάντων δεν είναι καταστροφή αν σε όλους τους τομείς έχουμε πάει στο 2%. Αυτά από ό,τι κατάλαβα όσον αφορά την κυκλική εναλλαγή των γενικών διευθυντών. Καταρχήν υπάρχουν κάποιοι κανόνε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάθε πενταετία, επταετία κυκλική εναλλαγή. Νομίζω ότι είναι ε, σωστό και εγώ στην ε, Κομισιόν άλλαξα πολλέ θέσει Δεν ε, κρίθηκε ότι θα πρέπει το να, αλλάξω καθήκοντα, οπότε έμεινα εκεί που ήμουνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντέλη. Ο Πρόεδρος. Για να κλείσουμε τώρα αυτό το σημείο τη διάταξη, τώρα θα δώσουμε τον λόγο στον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν θέλει. Κύριε Μουγκουρούθα, μας λέτε τις καταλητικές σας παρατηρήσεις από πλευράς συνεδρίου. Ο απλώς να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας. για τα όσα μας καλέσατε να πούμε. Του χρόνου στην εκθεσή μας θα επεκταθούμε στα θέματα αυτά της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στην κυκλική ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Έκλεισε επομένω και αυτό το τμήμα της ζήτησης Και τώρα θα συζητήσουμε τα της Όλαφ. Ποιος θέλει το λόγο. Αρχίζουμε το ΕΛΚ. Γκρέσλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσία και της ε, κυρίας Τεστόρη Κόζη. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, το ένα αφορά κάποια ζητήματα όπως το mail της 28 Σεπτεμβρίου 2012 της Γενικής Γραμματέως ε, όταν είχε ήδη ξεκινήσει η πρώτη υπόθεση και αφορά την αλλαγή της πρότασης οδηγίας για τα προϊόντα καπνού όπου λέγεται πως αναφέρονται κάποια αποτελέσματα και ακριβώς μιλάμε για, προϊόντα, για άκαπνα προϊόντα καπνού, δηλαδή συγκεκριμένα το σνούς, τα οποία θέλουν να μπουν στο, ε, στην οδηγία και από ό,τι φαίνεται ζητήθηκαν κάποια λεφτά το ερώτημα λοιπόν είναι τι γίνεται με αυτό εδώ το email. Ξέρουμε πως η κυρία Ντέι είναι πάρα πολύ προσεκτική και μας προξένησε σε έκπληξη η παρέμβαση αυτή στην διαδικασία ε, ε, λήψης αποφάσεων του Όλαφ. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, κάποια άλλα ζητήματα που φαίνεται πως οδηγούν σε μια λογική σαλαμοποίηση, δηλαδή τι ήξερε η Κομισιόν για τις μομφές της Swedish Match, πως επίτροπος ζήτησε λεφτά για να αλλάξει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στο πρώτο ερωτηματολόγιο, στη σελίδα, στην ερώτηση 20, λέγεται πως ε, πρόκειτο για κάτι το οποίο έφτασε απευθεία στη Γενική Γραμματέα από τη Swedish Match και μετά λέγεται πως ο κύριος Πετίτ τηλεφώνησε στην Γενική Γραμματέα και μετά επαναλαμβάνεται αυτό και στο τρίτο ερωτηματολόγιο στην ε, ερώτηση 29. Οπότε μας ενδιαφέρει η συνομιλία της κυρίας Ντέι και του κυρίου Πετίτ το τηλεφώνημα, αν μπορείτε να μας πείτε το τι διημήθη εκεί πέρα. Όσον αφορά επίσης τις επαφές υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας και της, υπηρεσ... της ε, νομικής υπηρεσίας. και από ό,τι φαίνεται φτάσαμε στα ανώτατα κλιμάκια και είχαμε και μία συνομιλία με τον ε, διευθυντή της νομικής υπηρεσίας. Οπότε πρώτα το email και δεύτερον γιατί λάβαμε διαφορετικές απαντήσεις στο ερώτημα για το πώς απευθύνθηκε η Swedish Match στην Γενική Γραμματεία. Ευχαριστώ. Οι Σοσιαλδημοκράτης τώρα ποιος θέλει το λόγο. Κανείς από ό,τι φαίνεται. Ούτε πράσινη. Α, ναι, παρακαλώ. Ναι, έχω κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα προς την κυρία Τεστόρη. Κυρία Τεστόρη, ως Γενική Διευθύντρια της ε, Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, ε, συνεργάζεστε με τον Επιτροπό Ντελή. στο διάστημα που συνεργαστήκατε σε αυτή τη θητεία υπήρξε κάποια στιγμή κατά την οποία σκεφτήκατε ο κύριος Νταλή εδώ πέρα προσπαθεί να δώσει κάποια κατεύθυνση στην ε, οδηγία αυτή που δεν συμφωνεί με αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Γενική Διεύθυνση. Είχατε ποτέ την αίσθηση πως ο κύριος Νταλή ή το περιβάλλον του προσπάθησαν να περιγράψουν το σνούς αυτό το προϊόν της Swedish Match με τρόπο ώστε να αλλάξει η νομοθεσία. Μετά η κυρία Γκρέσλε αναφέρθηκε στο email σας της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 προς την Catherine Day όπου μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των δικών σας υπηρεσιών και της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν καταλήξατε στο ότι το αρχικό κείμενο της οδηγίας προσαρμόστηκε σε έξι σημεία και τα έξι σημεία αφορούν προϊόντα ε, που μοιάζουν πάρα πολύ με τα προϊόντα της Swedish Match. Και προς την κυρία Day Αντιλαμβάνομαι πως ο ρόλος σας ως ε, Γενική Γραμματέας είναι να δώσετε μια καθοδήγηση στην διοίκηση να προσαρμόζονται οι κανόνες, να στέκουν νομικά τα όσα γίνονται, αλλά αντιλαμβάνομαι από όλη την αλληλογραφία και ηλεκτρονική αλληλογραφία που έχουμε τώρα, πως επίσης ε, μπαίνεται και στην πολιτική ε, διαμόρφωση των αποφάσεων και κατευθύνεται την πολιτική. Το ίδιο και για την οδηγία του καπνού και για την άλλη νομοθεσία έχω την εντύπωση πως ε, συμπεριφέρεστε ως ο 29ος ή 29η υπερεπίτροπος. Αυτή είναι η δουλειά σας. Πώς έχετε τόση δύναμη ώστε να κατευθύνετε το που θα πάει η νομοθεσία. Als nächstes hat sich jetzt noch gemeldet Sigmantas. Ο κύριος Σιγμάντας Μπαλτσίτης κατόπιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κι εγώ μία ερώτηση προς την κυρία Γενική σε σχέση με την οδηγία των πρώτων καπνών. Όπως ξέρετε μέχρι πρόσφατα είχαμε την προηγουμένη πρόεδρια του Συμβουλίου οπότε και βάλαμε εμείς το λιθαράκι μας σε αυτή την ε, δύσκολη οδηγία. Γνωρίζουν οι συναδελφοί βουλευτές ότι κάποιες καπνοβιομηχανίες έπρεπε να επενδύσουν πάνω από 100 εκατομμύρια για να προσαρμοστούν. Και ο κ. Βιτάτης Ζωκάκης ασχολήθηκε με αυτό. Άρα, Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάνουμε την μπορούσαμε για να προσαρμοστούμε και τώρα θέλω να ρωτήσω τον, ε, την κυρία Γενικό. Πρόκειται να κάνετε κάτι όσον αφορά τις σχέσεις ε, των λόμπι με τους βουλευτές. Γιατί είχαμε θέματα τέτοια ε, για την εν λόγω οδηγία, δεν πρέπει να τα κάνουμε. να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τις περιπτώσεις ε, συγκρούσεων συμφερόντων. Πρόεδρος. Και τώρα. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε την κυρία Πάολα, το της, την οποία καλώς ορίζω. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω ποια θέλει να απαντήσει πρώτη. Mrs. Day, please. Η κυρία Ντέι. Ναι, φαίνεται πως περισσότερες ερωτήσεις απευθύνονται σε μένα. Θα απαντήσω εγώ και μετά η συνάδελφος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυρία Γκρέσλι αναφέρεται σε διαφορετικές εκδοχές, γιατί η Κομισιόν έχει εξηγήσει επανειλημμένα το τι συνέβη. Και από γνωρίζω, εμείς πάντα την ίδια απάντηση δίνουμε, την αλήθεια. Η όλη αυτή η υπόθεση που αφορά τον Επίτροπο τον κύριο Ντάλη ξεκίνησε όταν έλαβα τηλεφώνημα από τον πρώην συνάδελφο, τον Μισελ Πετή, που είπε πώς τον προσέγγισε η Swedish Match με, μία, με έναν ισχυρισμό και ήθελα να μάθουν πώς θα ενημερώσουν την Κομισιόν. Του είπα λοιπόν πως εάν ήθελα να ενημερώσουν την Κομισιόν πρέπει να απευθυνθούν σε μένα που είμαι η Γενική Γραμματέας, εγώ, η Γενική Γραμματέας, με συγχωρείτε, εγώ είμαι το σημείο επαφής και αυτό του είπα και αυτή ήταν η μόνη επαφή που είχαμε. Το έχουμε πει επανειλημμένος, γραπτός, γιατί αυτό συνέβη. Όσον αφορά το email θα απαντήσουμε και εγώ και η Πάολα, αλλά θα ήθελα να απαντήσω και στο ερώτημα του κυρίου Στάς για τον ρόλο μου στην Κομισιόν. Ο ρόλος μου περιγράφεται σε μια επίσημη απόφαση της Κομισιόν για τις 15 Νοεμβρίου ε, στις 15 Νοεμβρίου 2005 προφανώς κανείς δεν φανταζόταν γυναίκα ε, γιατί λέει συνεχώς ο Γενικός Γραμματέας αλλά ε, εγώ το ερμηνεύω ότι μπορεί να αφορά και γυναίκες και λέει πως ο Γενικός Γραμματέας προετοιμάζει τη διεξαγωγή των ε, συναντήσεων και λέει μετά ο Γενικός Γραμματέας θα, θα βοηθά στο συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 23 και θα φροντίζει πως τα έγγραφα που υποβάλλονται στην Κομισιόν είναι επαρκούς ποιότητας και σύμφωνα με τους κανόνες και στο άρθρο 23 λέει πως η Γενική Γραμματεία θα ενημερώνεται για όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν πολιτική σημασία, που αποτελούν μέρος του ετησίου προγράμματος εργασίας της Κομισιόν ή αφορούν θεσμικά ζητήματα ή ε, είναι αντικείμενα διαβούλευσης ή μελετών αντικτύπου. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό κάνω και αυτό σημαίνει πως και η Γενική Γραμματεία και η Νομική Υπηρεσία παίζουν τον κανονικό τους ρόλο στην προετοιμασία των ε, ε, διαφόρων μοθημάτων όπως και στην οδηγία για τα προϊόντα καπνού και θα έλεγα πως πράγματι η νομική υπηρεσία πρέπει να λέει τη γνώμη της για όλα τα νομικά έγγραφα. Εδώ πέρα λοιπόν είχαμε μια νομοθετική πρωτοβουλία. Ε, είχε απορριφθεί από το δικαστήριο προηγούμενη πρόταση της Κομισιόν γιατί θεωρούσε πως η Κομισιόν είχε υπερβεί τη νομική βάση. Οπότε δεν υπάρχει κανένα μυστήριο εδώ πέρα, έτσι λειτουργεί η Κομισιόν. Έχουμε 28 επιτρόπους, 30.000 υπαλλήλου, πολλά πράγματα πολλά πράγματα τρέχουν παράλληλα. Υπάρχει η εντολή μας για τον συντονισμό και εντό αυτού του πλαισίου λειτουργώ ως υπάλληλο και μόνο ως υπάλληλο. Για το ζήτημα του email θα απαντήσει και η Πάολα αλλά το email το οποίο αναφέρατε απλά ήταν μέρος αυτής της διαδικασίας εσωτερικών διαβουλεύσεων για το τι είναι νομικά δυνατόν όσον αφορά τις δραστηριότητες στον τομέα της υγείας αλλά και το ότι η Κομισιόν είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της ε, να ε, ληφθούν υπόψη ε, πράγματα όπως η αξιολόγηση, η δημόσια διαβούλευση κτλ. Αν συμφωνείτε τώρα θα δώσω λόγο στην συνάδελφό μου για τις ερωτήσεις που την αφορούν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Στάς που έθεσε τα δύο αυτά ερωτήματα. Απαντώ στο πρώτο. Και ουσιαστικά εδώ πέρα λέω τα ίδια πράγματα που είπα και στην ε, Όλαφ όταν χρειάστηκε να κάνω μια δήλωση κατά την έρευνα που έγινε για τον κύριο Ντάλι. Σε καμία περίπτωση δεν είχα την εντύπωση ότι ο κύριος Ντάλι προσπάθησε να υπονομεύσει την πρόταση αυτή για την οποία εργαζόταν η γενική μου διεύθυνση. Το ζήτημα του σνούς που είναι ένα από τα αμφιλεγόμενα ζητήματα ανέκαθεν ναι, αντιμετωπίστηκε με την ίδια στάση, με την ίδια προσέγγιση. Θέλαμε εμεί να διατηρήσουμε του ίδιου κανόνε για το σνούς. Ουδέποτε λοιπόν συζητήσαμε αν θα πρέπει να απελευθερωθεί όχι το συγκεκριμένο προϊόν καπνού. Αυτό για το πρώτο σα ερώτημα. Το δεύτερο που έχει να κάνει και με αυτά που είπε η κυρία Γκρέσλερ για το mail αυτό τη 7 η Σεπτεμβρίου. Στο email αυτό, το οποίο αναφέρεται σε μια συζήτηση που είχα με τους εργαζομένους μου από την Γενική Διεύθυνση καθώς επίσης και από την Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν το τελευταίο στάδιο μίας διαδικασίας μακράς που ξεκίνησε το 2009. Ας μην ξεχνάμε ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού ξεκίνησε το 2009 και όλες οι εξολογήσεις αντικτύπου επιταχύνθηκαν το 2011 και το 2012. Αν δούμε λοιπόν την ουσία, τα τρία σημεία, έξι συνολικά είναι. Υπάρχουν πάντως τρία σημεία για τα οποία θα έλεγα ότι μπορείτε να πείτε ότι εσείς, θα μπορείτε να πείτε εσείς ότι εγώ συμφωνούσα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν τρία σημεία για τα οποία συμφώνησα να γίνουν κάποιες αλλαγές και ουσιαστικά να καταστήσουμε κάπως πιο ήπιους τους κανόνες που προτείνονται. Ουσιαστικά δεν αποφασίζαμε εκείνη τη στιγμή για μια γενική απαγόρευση των προϊόντων καπνού, γιατί αρχικά θέλαμε να απαγορεύσουμε όλα τα... Όλα τα προϊόντα αυτά καπνού, τα άκαπνα όπως το σνούς. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση που είχε γίνει. Αποφασίσαμε όμως να μην απαγορεύσουμε τις άλλες μορφές προϊόντων καπνού, τον καπνό που μασάμε κτλ. Γιατί είχε γίνει μια πολύ εκτενή συζήτηση στη νομική υπηρεσία και είδαμε ότι ήταν δύσκολο αν χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 114 της συνθήκης να καταφέρουμε να δικαιολογήσουμε μία ολοκληρωτική απαγόρευση. Με το άρθρο 114 μπορεί κανείς να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά την χρήση, την πώληση, την ετικετοθεσία, αλλά δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να βασιστούμε στο άρθρο αυτό και να προχωρήσουμε σε πλήρη απαγόρευση. Ξέρετε, ξέρετε επίση ότι στην περίπτωση προσφυγών θα πρέπει να είμαστε σε θέση να υπεραμειθούμε τις τάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να νικήσουμε τη δίκη. Επίσης, ε, γίνανε κάποιες άλλες εικασίες για το ότι ε, εγκαταλείπαμε τους ε, αρχικούς κανόνες που υπήρχαν όσον αφορά τις μηχανές αυτόματης πώληση των προϊόντων αυτών. Και πάλι εδώ πέρα θεωρήσαμε ότι δεν υπήρχε λόγος να νομοθετήσουμε για κάτι το οποίο διευθετείται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και μας είπατε επίσης ότι εγκαταλείπαμε την όλη ιδέα της απλής συσκευασία, γιατί αρχικά η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ήθελε να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να επιλέξουν την απλή συσκευασία, αλλά ήθελε επίσης και να αρμονιστεί η απλή συσκευασία. Εμείς εγκαταλείψαμε λοιπόν την ιδέα αυτή για την νομική υπηρεσία κατέδειξε ότι ήταν πολύ πιο εύκολο να πούμε ότι ό,τι δεν ρυθμίζεται παραμένει ως έχει, δηλαδή ένα 25% της επιφάνειας συσκευασίας θα αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όλες αυτές λοιπόν οι τρεις αλλαγές δεν υπονομεύουν, δεν αποδυναμώνουν την οδηγία. Και αυτό ακριβώς προσπάθησα να αποδείξω τώρα. για τα σημεία αυτά και κυρίως για το πρώτο σημείο, δηλαδή η ρύθμιση όσον αφορά τα στατικά των προϊόντων καπνού, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποδυνάμωσαν πολύ περισσότερο τα ίδια τη δική μας αρχική πρόταση. Σας το λέω αυτό για να σας πω ότι η δική μας η πρόταση ήταν πιο φιλόδοξη από αυτή που τελικά προτάθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Okay, uh, Και άλλοι συνάδελφοι τώρα έχουν ζητήσει το λόγο. Ως πρόεδρος, θέλω να πω το εξής. Σχολήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με το θέμα από τις αποχώρησεις του κ. Ντάλη και υποβάλαμε κάποιες ερωτήσεις και δεν λάβαμε απαντήσεις. Ή τέλο πάντων ε, οι απαντήσεις που λάβαμε δεν μας κάλυψαν. Η δε διάσκεψη των Πρόεδρων του Κοινοβουλίου απεφάσισε να καλέσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, του κύριο Μπάουσο. Και έτσι θα συνομιλήσουμε μαζί του. Όμως, δεν υλοποιήθηκε η απόφαση αυτή. Στη συνέχεια αποφάσισε η Διεύθυνση των Πρόεδρων ότι εμείς έχουμε την αρμοδιότητα του να υποβάλουμε σχετικές ερωτήσεις. Πολλές φορέ με τις επιστολές αυτές που ανταλλάσσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει την εντύπωση ότι. Ε, έστω και υποκειμενική εντύπωση δημιουργείται ότι υπάρχει. υπάρχει έλλειψη κατανόηση του γιατί τι θα διαρωτήσω όμω, νομίζω σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία ο κοινοβουλευτικό ε, δημόσιο έλεγχο, ε, ο έλεγχο ε, επί τη εκτελεστική εξουσία, είναι κάτι το επιβαλλόμενο και επομένω δεν πρόκειται για προσωπικό ψόγο και άλλωστε είμαστε κοινοβούλιο άμεσα εκλεγμένο. Οπότε είναι θεμητή υποβολή αυτών των ερωτημάτων σε σχέση με την ε, υπόθεση Ντάλι. Κύριε έχω κάποια ερώτηση. Υπάρχουν κάποια σημεία ιδιότυπα. Αν πάρετε δε κάποιες πληροφορίες, αν έχετε πληροφορίε από την όλα όσον αφορά την υπόθεση αυτή της δωροδοκίας, θεωρείτε ότι υπάρχει μηχανός προστασία επαρκή για να προστατεύσει τους ε, επιτρόπους από πλευράς διοικητική. Γιατί εάν κάποιο ε, λόμπι προσεγγίσει κάποιον ε, υψηλόθωμο υπάλληλο, κάποιον επίτροπο, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος προστασίας από κάποιο μηχανισμό, από κάποιο πλέγμα διατάξεων. Εσείς, τι θεωρείτε, ότι υπαρκεί το ισχύον πλαίσιο ή θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Και αν δεν μπορείτε να απαντήσετε ευθύ αμέσω, τότε με ικανοποιεί και γραπτή σα απάντηση. Τώρα οι άλλοι συναδελφοί που θέλουν να λαβούν το λόγο. Κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς και απευθύνομαι στην κυρία Ντεΐ. Κοιτάξτε, ξέρουμε πως 8 και 9 Μαΐου ο κύριος Πετή, ως εκπρόσωπος ε, μιας καπνοβιομηχανίας, σας τηλεφώνησε. Γιατί είπατε στείλτε μας εμάς, να το στείλει σε εμάς η Swedish Match, ενώ κανονικά θα ήταν περίπτωση Όλαφ. Και όταν αντιμετωπίζει κανείς μια τέτοια μομφή προσπαθεί να απομακρυνθεί από ένα τέτοιο ζήτημα γιατί είναι μια προβληματική ε, ιστορία γιατί λοιπόν να πάει αυτή η καταγγελία στην Γενική Γραμματέα. Και τι είπατε, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω. Μετά, η περίπτωση στην έχει πάρα πολλές πτυχές. Είδαμε πως ε, στις 27 Μαρτίου ήδη υπήρχε μία συνάντηση με τον κύριο Φεριέ, με τη Γενική ε, γραμματεία και υπάρχει αυτή η ένωση σνούς που έπαιξε ένα ρόλο και δεν συζητήθηκε από ό,τι φαίνεται η κατηγορία η οποία ήδη υπήρχε και μετά 21 έκτου υπήρξε μια συζήτηση μεταξύ του γραφείου του Μπαρόζο και πάλι αυτού του συνδέσμου για το σνούς. Θα ήταν κάπως περίεργο δηλαδή ένας σύνδεσμος που κάνει μια τέτοια μομφή εις βάρος επιτρόπου να μην το συζητήσει το θέμα αυτό με τον κύριο Μπαρόζο. Επίσης αν θα μπορούσαμε να έχουμε τα πρακτικά της 27ης ε, Τρίτου και 21ης ε, Ιουνίου 2012 θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Μετά το ζήτημα το ερώτημα που δεν απαντήθηκε, οι, ερωτήσεις με τον, οι συναντήσεις με τον κύριο Πετίτ και η επαφή με τους υπαλλήλους νομικής υπηρεσίας. Στην απάντηση 15, στο πρώτο ερωτηματολόγιο, μιλάτε για επαφές και μάλιστα υπήρχε μια επαφή το Σεπτέμβριο του 2012 με τον κύριο Πάτρικ Χέτζ και τον Μάρκ Φανχόφ ε, Σεπτέμβριο του 2012. Και υπενθυμίζω πως οι επαφές αυτές γίνονταν πάντα όταν είχαμε μία νέα φάση της οδηγίας καπνού. Δηλαδή, Σεπτέμβριο είχαμε την αξιολόγηση αντικτύπου και μετά, πριν από την ε, εσωτερική συνεννόηση, είχαμε μετά, ήταν ακριβώς μετά την ε, αξιολόγηση αντικτύπου. Φοβερές συμπτώσει, δηλαδή. Ε, θα ήθελα να μάθω τι άποψη έχετε κύριε Αντέ, γιατί έχουμε πραγματικά φοβερή πρόσβαση στις εσωτερικές διαδικασίες της Κομισιόν. Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν τηλέφωνο, να σας μιλήσουν σε κάθε φάση μιας εσωτερικής διαδικασίας, για την οποία φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλά πληροφορημένοι γιατί νομίζω και ο κ. Φέτς ήταν ε, ε, αναπληρωτής διευθυντής της νομικής υπηρεσίας ε, και ο άλλος ήταν ε, συντονιστής της διαδικασίας για την οδηγία καπνού. Για την κυρία Τεστόρικο, αυτά που γράψατε μας είπατε, πράγματι. Εγώ θεώρησα πως ήταν πάρα πολύ καλή πρόταση, αλλά για ένα πράγμα δεν μας είπατε κάτι για την αναβολή της πρότασης. Γιατί η πρόταση αναβλήθηκε. Και συμφωνώ εδώ πέρα μαζί σας. Δεν έχω καταλάβει μέχρι σήμερα πώς ε, δεν επιτρέπεται να φτάσει αυτή η πρόταση, δεν επιτράπηκε να φτάσει στους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Μπαρτ Στάς. θα αναφερθώ και εγώ σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκρέσλε. Αναφέρθηκε στις επαφές ε, του κυρίου Πετίτ με τον Πάτρικ Χέτς το Σεπτέμβριο του 2012 και τον Μάρκ Φανχόφ ε, επίσης. Αλλά στις 14 Νοεμβρίου 2012 υπήρχε μια συνάντηση μεταξύ ε, Πετίτ και του κυρίου Ρομέρο, διευθυντή της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου τι συζητήθηκε εκεί, γιατί πρέπει ένας ε, δικηγόρος ε, επιχειρήσεων, πρώην υπάλληλο ε, της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν, τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται μας είπε η κυρία Τεστόρη είχαμε μια τελική συμφωνία μεταξύ της DG Sanko και νομικής υπηρεσίας και μας είπε τα τρία από τα έξι σημεία κυρία Τεστόρη, γιατί πρέπει να υπάρξει μια χωριστή συνάντηση 14 Νοεμβρίου 2012 με έναν λομπίστα, έτσι, εκπρόσωπο της καπνοβιομηχανίας και του διευθυντή της νομικής υπηρεσίας. Έτσι. Αξιοσημείωτο. Αυτό το οποίο επίσης βρίσκω περίεργο είναι πως όταν ε, φτάσαμε σε τελική συμφωνία DG Sanko και νομικής υπηρεσίας και άρα επιτέλους δεν υπήρχαν άλλα εμπόδια για να ξεκινήσει η κανονική εσωτερική διαδικασία και όλα από ό,τι φαίνεται ήταν έτοιμα μέσα Σεπτεμβρίου από ό,τι φαίνεται από τα email γιατί αναβάλλεται συνεχώς αυτή η εσωτερική συνεννόηση των υπηρεσιών της Κομισιόν και η κυρία Τεστόρη ζητάει να επιταχυνθεί η διαδικασία, η κυρία Ντέι το αρνείται και θέλει να αναβληθεί μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των αρχών Οκτωβρίου. Εντάξει, είναι ευαίσθητα τα πράγματα και μας λέτε εδώ πέρα πως δεν θέλω να τα επηρεάσει αρνητικά το Συμβούλιο τα του Καπνού, μα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφορούσε την Ευρωκρίση, έτσι είχε σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί. Δεν νομίζω να το απασχολούσε η οδηγία του Καπνού και να την επηρεάσει αρνητικά και επιπλέον λαμβάνει χώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπάρχει έτοιμα μετά να ξαναξεκινήσει η εσωτερική συνεννόηση και αναβάλλεται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Αρχές Δεκεμβρίου 2012. Και μετά πάει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι είχα, είχε γίνει η προετοιμασία, κινούνται τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε το ερώτημα είναι το πώς ε, ζητάει η κυρία Νοεμβρίου να μην γίνει πάλι η συνεννόηση 11 Νοεμβρίου, ε, ε, Δεκεμβρίου, με αλλά 19 Δεκεμβρίου για να ξαναπεράσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μα τι σχέση έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων με την εσωτερική συνεννόηση των υπηρεσιών ή των 28 επιτρόπων για μια πρόταση ε, οδηγίας. Δεν το καταλαβαίνω. Αν μπορείτε να μου το εξηγήσετε, ποιο είναι το σκεπτικό σας εδώ πέρα, που λένε και στα αγγλικά. Ναι, σας ευχαριστώ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Παρακαλώ να μας απαντήσετε. Thank you very much. Um, Mr. Chairman, let me... Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι σε σχέση κάτι που είπατε Εσεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με καμία έννοια δεν διαφωνεί με το ότι πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτικό δημόσιο έλεγχο. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά Εσεί δεν είστε 100% ικανοποιημένοι όπως το είπατε και αυτό διότι σε κάποιες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Πρόκειψε ότι εμεί θα πρέπει να σεβαστούμε το ότι και αυτή η, υπόθεση εκκρεμωδική ακόμα σε κάποια κρατημέλη. Βεβαίω και πρέπει να σα εξηγήσουμε τι έχει γίνει. Αλλά όμω από την άλλη μεριά, εκτό από την υποχρέωση να σα δώσουμε λόγο, θα πρέπει να σεβαστούμε την εκκρεμωδική. Μα ρωτήσατε κάτι για την Όλαφ. Δεν είναι δικό μα αρμοδιότητα. Απάντησε η Όλαφ για τα τη Όλαφ. Πάντως, Σα είπαμε να σας πούμε εκτενώ. Αυτό ελπίζω σας καθησυχάσει. Επίσης, ρωτήσατε αν χρειάζεται προστασία η Επίτροπη. Υπάρχει κώδικα διοντολογία για τους επιτρόπους. Ορίζει τι πρέπει να κάνουν. Επίση, έχουμε το πρωτόκολλο διαφάνειας κοινό μαζί σας. Εκεί εκουσίω έχουν καταγραφεί, εγγραφεί χιλιάδες λομπιστών. Μην είναι σαφές για αυτούς που θέλουν να τους τους επιτρόπους. Θα πρέπει όποτε έρχονται σε επαφή με επίτροπο να είναι ξεκάθαρο το τι θέλουν. Μην έχουμε πολυνομία. Δεν είμαστε τόσοι πολλοί επίτροποι σε σχέση με την ύλη μας. Οπότε χρειαζόμαστε κάποιες συμβουλές. Είμαστε ανοιχτός οργανισμός. Πολύ πιο ανοιχτό από τι εθνικέ κυβερνήσει. Όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να μάθει τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Άρα αυτό το ανοιχτό πνεύμα, η ανοιχτή φύση θα πρέπει να συμβάζεται με την διαφάνεια και με το ότι πρέπει να ακούμε όλες τις απόψεις. Θέλουμε να μιλούμε με αντιπροσωπευτικούς φορείς, φορείς που έχουν τους διαφορούς κλάδους. Τώρα για τους νέους κανόνες, όταν έρθει η θητεία της νέας Κομισιόν, θα προσπαθήσουμε να τους εξοικειώσουμε, τους καινούριου με το ισχύον πλαίσιο. Επομένω είναι θέμα κατανόηση, θέμα εξισορρόπηση. Να μην επηρεαζόμαστε από τις ομάδε πίεση και ταυτόχρονα είμαστε ανοιχτοί. Ε, κύριε Γκρέσλε, σε σχέση με την τηλεφωνική μου αυτή επαφή. και το πώς προσύγγισε η εταιρεία αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός ο ισχυρισμό σοκάρει. Αφορά επίτροπο. Αν υπάρχουν ισχυρισμοί για αδόκιμη συμπεριφορά θα πρέπει αυτό να διατυπωθεί επισήμως. Διατυπώθηκε επισήμως και παρεπέμφθη το ζήτημα ή στην αυτό όπω όφιλε. Δεν έχουμε κάτι άλλο όπως έχω πει και δηλώσει. Μόνο με τον κύριο Πετή ήταν αυτό το τηλεφώνημα. Του εξήγησα καθώς μια φορά. Και μου ζήτησε συμβουλή και εγώ τη συνεβούλευσα και είπα ότι όλα θα πρέπει να πρωτοκολληθούν και να γίνουν όπως πρέπει. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει στην Επιτροπή. Επίσης, αποκαλύψαμε κάθε επαφή, κάθε πληροφορία, ό,τι επαφές είχε η Επιτροπή σε σχέση με την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Καλά, δεν είναι καταγεγραμμένες όλες οι συναντήσεις, αλλά υπάρχουν όσα υπάρχουν. Έχουμε απαντήσει στα υπόλοιπα, δεν έχουμε προσθέσει τίποτα άλλο. Γιατί αναβλήθηκε τώρα η εισήγηση στη, στο σώμα των Επιτρόπων. Έχουμε τις διατάξεις σε σχέση με την οργάνωση της Επιτροπής και το ρόλο του Γενικού Γραμματέα, η Επιτροπή καταρτίζει την μέση διάταξη ανάλογα με τα θέματα, τον διαθέσιμο χρόνο. Και θα έπρεπε ταυτόχρονα με τις αντίσεις του Προέδρου με το Συμβουλίο έπρεπε να κάποιο, να συζητήσει κάποια τρέχοντα θέματα. Η αναβολή δεν γίνεται κάθε μέρα, αλλά γίνεται αρκετά συχνά, ανάλογα με τις ανάγκες. Ανάλογα με το αν ενδιαφέρεται το κοινοβούλιο, ανάλογα εάν ε, βοηθάει την φραγμός εργασία του Συμβουλίου. Μιλάμε για 28 πρόσωπα. Έχουν τόσο πολλά να κάνουν πρέπει να οργανώνονται συνεδριάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε τα θέματα να έρχονται προς συζήτηση όταν μπορούν οι επιτροποί με σοβαρότερα να τα συζητήσουν. Ο κανομοθέτημα που απαιτεί συζήτηση. Προετοιμασία, ας πούμε, για το MFF. Είπαμε ότι θα διτυπώσουμε κάποια πρόταση. Κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα με τη σειρά μου. Για το σημείο αυτό, ο κύριος Στάς μας είπε κάποια πράγματα και όντω εγώ είχα επαφές με τη Γενική Γραμματέα και με την Νομική Υπηρεσία σε αρχές Σεπτεμβρίου στη συζήτηση αυτή. Μιλήσαμε για τα τελευταία στοιχεία που είχαμε σε σχέση με την πρόταση αυτή και χρειάστηκε όλος ο μήνας Σεπτέμβριος για να ολοκληρωθεί το έγγραφο αυτό και έπρεπε από νομικής πλευράς να ελέγξουμε ουσιαστικά το κείμενο και στα τέλη Σεπτεμβρίου η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ υπό τη δική μου την επιτήρηση άρχισε να ασκεί πίεση προκειμένου να εγκριθεί το κείμενο αυτό πριν τα Χριστούγεννα, γιατί η Κυπριακή Προεδρία δεν θα ξεκινούσε τη συζήτηση γιατί δεν ενδιαφερόταν για το ζήτημα αυτό. Θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε η Ιρλανδική Προεδρία γρήγορα να ασχοληθεί και να εγκρίνει την πρόταση αυτή. Εμεί είπαμε ότι πριν τα Χριστούγεννα θέλαμε να εγκριθεί το κείμενο. Όταν το συζητήσαμε με την Κάθριν και είπε τότε ότι ήταν καλύτερα να περιμένουμε τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια εντελώ αναμενόμενη αντίδραση. Είναι πολύ σημαντικό όταν ξεκινάνε οι διοργανικέ διαπραγματεύσει να συζητάμε με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Αυτό κάνουμε για κάθε ζήτημα άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το ακόλουθο. Μετά την αποχώρηση του κυρίου Ντάλη στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ συνειδητοποίησαμε ότι δεν θα ήταν δυνατό να έχουμε τη διοργανική διαπραγμάτευση και έγκριση του κειμένου αυτού χωρίς να έχουμε έναν αρμόδιο επίτροπο. Επομένως σταματήσαμε να ασκούμε πίεση, συνεχίσαμε να εργαζόμαστε με την νομική υπηρεσία προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι μεταφράσεις έτσι ώστε αυτή τη στιγμή θα αναλάμβανε τις υποχρεώσεις του ο νέος αρμόδος επίτροπος θα μπορούσαμε γρήγορα να ξεκινούσαμε τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, πράγμα το οποίο και έγινε. Στον Επίτροπο Μπόρκ έστειλε μια επιστολή 28 Νοεμβρίου για να ξεκινήσουν οι διοργανικέ διαπραγματεύσει, αμέσω συμφώνησε την επόμενη μέρα στι 29 ο κύριο Μπόρκ. Ξεκίνησε η διοργανική διαπραγμάτευση ή γίνανε όλε οι μεταφράσεις και καταφέραμε σε χρόνο ρεκόρ να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Μετά από αίτημα λοιπόν τη Γενική Διεύθυνση ΑΝΚΟ για έγκριση πριν από τα Χριστούγεννα καταφέραμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα αυτό το φάκελο. Yeah, Σας ευχαριστούμε πολύ, ο κύριο Στάσπάλι. Καταλαβαίνω την απάντηση της κυρίας Ντέι. Εντάξει, καταλαβαίνω να υπάρξει μία αναβολή κάποιων θεμάτων λόγω της πολιτικής ατζέντα και το ότι θα είναι δύσκολες οι συζητήσεις σε μία συνεδρίαση των ε, επιτρόπων όπου θα συζητηθούν πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Το καταλαβαίνω αυτό, έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ανεξαρτήτως ε, της ε, απόλυσης του κυρίου Νταλή, αλλά η κυρία Τεστόρη λέει πως ε, εντάξει δεν ξεκίνησε η εσωτερική συνεννόηση τον Οκτώβριο γιατί ο κύριος Νταλή αναγκάστηκε να παρετηθεί αλλά αυτό δεν εξηγεί και δεν μας εξηγήσατε κυρία Ντέι το γιατί συνδέεται η έναρξη της εσωτερικής διαδικασίας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Δηλαδή, τι σχέση έχει το ότι 28 πρωθυπουργοί θα συναντηθούν με ε, το εάν ε, θα συνεννοηθούν μεταξύ τους οι υπηρεσίες κομισιών. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. ναι, σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Να επανέλθω λίγο. Λέτε πως το πρωτόκολλο των συναντήσεων μεταξύ των εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας ε, και του γραφείου του κυρίου Μπαρόζο δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν πρακτικά αλλά υπάρχουν οι κατευθυντήριες γραμμές ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ε, που λένε πως ε, πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα, δηλαδή πρέπει να τηρούνται πρακτικά όταν συναντάει κανείς εκπροσώπους καπνοβιομηχανίας. Πώς το εξηγείτε λοιπόν αυτό όταν συναντάει η Σάνκο τους λομπίστες στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού δεν υπάρχει διαφάνεια. Προξένει προξένησε έκπληξη, όπως είπα, ε, το πώς πολλές επαφές υπήρχαν μεταξύ των υπαλλήλων της Κομισιόν και των υπαλλήλων καπνοβιομηχανιών σε όλα τα επίπεδα. Κατόπιν, ένα άλλο ερώτημα. Ρωτήσαμε πάντα, με τι σχέση έχει η συμφωνία του καπνού με την υπόθεση του Όλαφ. Εκεί πέρα βλέπουμε πως υπάρχει μία ρήτρα για πιθανή αυστηροποίηση της ε, νομοθεσίας ε, αυτής. Και όλοι όσοι ήταν στις διαπραγματεύσεις ε, μας είπαν πως ήταν όρος απαράβατος, πως δεν θα πρέπει να αυστηροποιηθεί η οδηγία περί προϊόντων καπνού. Τώρα όμως το 2015 εκπνέει η πρώτη συμφωνία με τη Φίλιπ Μόρις ε, που είχαμε και τις σχετικές πληρωμές. Ποιες δυνατότητες υπάρχουν λοιπόν για παράταση αυτής της συμφωνίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ντέι. Ευχαριστώ να σας εξηγήσω για άλλη μια φορά για ποιο λόγο διαχειρίστηκε έτσι τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την πρόταση αυτή για την οδηγία και σε σχέση με άλλα πράγματα τα οποία εξελίσσονταν παράλληλα εκείνη την περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ή άλλα ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ουσιαστικά να επικεντρώσει το ενδιαφέρον στα ζητήματα τα οποία βρίσκονται προς συζήτηση. Αν είχαμε ξεκινήσει λοιπόν την διυπηρεσιακή αυτή συζήτηση για την οδηγία προϊόντων καπνού παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τότε πραγματικά θα είχαμε πάρα, πολλές, πάρα πολλά αιτήματα συζήτησης για διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ουσιαστικά θα μονοπολούσαμε εμείς μέσω της ε, διπηρεσιακής αυτής συζήτησης την ίδια την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μολονότι το σώμα των επιτρόπων δεν θα έχει αρχίσει ακόμα επίσημα να συζητά τα ζητήματα αυτά και ενώ δεν θα μπορούσαμε ακόμα εμείς να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για τα υποσυζήτηση ζητήματα. και ιδίω ε, για δύσκολες συζητήσεις όπως για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε πραγματικά να τονίσει την γραμμή την οποία είχε οθετήσει. Έτσι λοιπόν εμείς δεν θέλαμε να αποπροσανατολιστεί όλη αυτή η ε, συζήτηση που έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει σοβαρά από άλλα ζητήματα τα οποία λάμβαναν χώρα και συζητώνταν εκείνη την περίοδο. Όπω είπε η επικεφαλή τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, είχαμε πει ότι μετά Χριστούγεννα θέλαμε να εγκριθεί οδηγία, πράγμα και το οποίο έγινε. Πολύ συχνά πάντω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε χώρε διαπραγματεύσει, διεθνεί διαπραγματεύσει, έχουμε ζητήματα τα οποία τελευταία στιγμή μα ζητά να διεκπαιρώσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να μην κάνουμε και αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και πρέπει κάθε φορά να δούμε πώ σχετίζονται τα ζητήματα τη ατζέντα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτά τα οποία συζητεί για παράδειγμα το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο και το πόσο ουσιαστικά επικεντρώνει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στο ένα ή στο άλλο ζήτημα. Και η Πάολα θα πάρει το λόγο να μιλήσει για τα ζητήματα αυτά σε λίγο. Ουδέποτε πάντως υπήρχε μία μυστική συμφωνία για το ότι δεν θα μπορούσαμε εμείς να πούμε συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά την οδηγία αυτή λόγω συμφωνίας που υπήρχε από το 2004. Η κυρία Τεστόρη Κότζη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει ένα non-paper για τα ζητήματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το οποίο, σύμφωνα με τη δική μας ερμηνεία, η θέση σε ισχύ της νέας αυτής οδηγίας για τα προϊόντα καπνού δεν θα επέτρεπε στους εκπρόσωπους της καπνοβιομηχανίας να ολοκληρώσουν, να τερματίσουν τη συμφωνία αυτή. Προβλέπονται κάποιες διατάξεις συμφωνία αυτή που θα συνεχίσουν να ισχύουν ανεξάρτητα από νέες οδηγίες ή προσαρμογές στην οδηγία που θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας θα συνέχιζε να ισχύει ούτως ή άλλως μετά την έγκριση της οδηγίας. Και άλλωστε όπως το είπατε προβλέπεται μία περίοδος από το 2016 στο 2029. Και νομίζω ότι οι σχετικές πληροφορίες έχουν δοθεί και άλλωστε Πρόεδρος. Κοιτάξτε. Πλησιάζει και το τέλος συνεδρίασης, αλλά κυρία Γκρέσλε έχει άλλη μια ερώτηση. Κυρία Ντέι ξέχασε την ερώτηση των πρακτικών της συνάντησης υπαλλήλων της Κομισιόν και δεν υπάρχουν από ό,τι φαίνεται πρακτικά παρά τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΗ. Και μετά επίσης την παράταση της ε, συμφωνίας. Ε, όπως είπε. Ευχαριστώ. Um, um, Μα νόμιζα ότι απάντησα στην ερώτησή σας για τα πρακτικά σε δύο συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις δεν είχαν διατηρηθεί τότε πρακτικά, αλλά νομίζω ότι ε, στο πλαίσιο του ε, Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προβλέπεται ότι για κάθε συνάντηση θα πρέπει να κρατώνται πρακτικά, επομένως θα ακολουθήσουμε και εμείς τη σύσταση αυτή. Τώρα δεν νομίζω ότι εκκρεμούν περαιτέρω διευκρινήσεις όσον αφορά την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Τα είχαμε πει όλα, Πρόεδρος. ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Έχω την εντύπωση πως θα μας απασχολήσουν κάποια από αυτά τα ζητήματα και στο μέλλον και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντέι και νομίζω καλό είναι να ξανασκεφτούν στο μέλλον πώς ε, μπορούν να προστατεύσουν επιτρόπους και στελέχη της ε, Κομισιόν γιατί δεν είναι δυνατόν ε, λομπιστές, λομπίστες να χρησιμοποιούνται για να ασχίσουν πίεση στην Κομισιόν στην προετοιμασία της νομοθετικής διαδικασίας. Πρέπει να σκεφτούμε επίσης πώς θα ενισχύσουμε την διαφάνεια και βεβαίως αυτό το οποίο θέλουμε όλοι μια καλύτερη προστασία από την διαφθορά. Σας ευχαριστώ. Διακόπτεται η συνεδρίαση και... Συνεχίζουμε στις 3 ώρα. Ευχαριστώ.